So, Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μέρα της ε, διήμερης ε, συνεδρίασής μας. Πρωτού περάσουμε στις πληροφορίες, επιτρέψτε μου σας παρακαλώ να σας δώσω κάποιες πληροφορίες σχετικά με την χθεσινή συνεδρίαση των συντονιστών της Επιτροπής Αναφορών. Μια τεχνική πληροφορία να σας δώσω, καταρχάς. Στις ε, 3.30 σήμερα το απόγευμα, το σημείο 31 θα ε, συζητηθεί πριν από το σημείο 30, το οποίο και θα συζητηθεί γύρω στις 4 το απόγευμα. Και τώρα κάποια γραφειοκρατικά θέματα. Με συγχωρείτε, αλλά είμαι υποχρεωμένος να, να σας ενημερώσω. Οι συντονιστές της ΠΕΤΗ αποφάσισαν χθες το απόγευμα τα εξή. Πρώτον, έγκριση της ημερήσια διάταξη Νοεμβρίου και αιτήματα για ε, μελλοντικέ ημερήσιε διατάξης. Ε, αναφορά 93-2017 θα προσθεθεί στην ημερήσια διάταξη του Ιανουαρίου. Η 1845 θα ε, ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη μετά την παραλαβή της απάντησης της Η 17 του, 2010, του 2012 σε σχέση με την ε, εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου θα προσθεθεί στην ημερήσια διάταξη αφού λάβουμε απάντηση από το, το Κοινοβούλιο της Σλοβακίας. Άλλα ζητήματα συνδέονται με συνεδρίαση 21 και 22 Νοεμβρίου. Εβδομάδα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Συμφωνήσαμε να ε, προσκαλέσουμε τον ύπατο ε, εκπρόσωπο της, ε, της ΥΠΑ της Αρμοστίας, τον, τον πρόεδρο της ΥΠΑ της Αρμοστίας ε, του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Επίσης θα γίνει ανταλλαγή απόψεων με τη Διαμεσολαβήτρια σχετικά με, την, με τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Κομισιόν στις 21 Νοεμβρίου στις 2.30 σε κοινή συνεδρίαση με τις Επιτροπές Γιούρι και Κοντ. Άλλα θέματα. Συμφώνησαν οι συντονιστές, ο πρόεδρος, να προσκαλέσει ε, η Κομισιόν αναφέροντες στο κολόκουιουμ για τα θεμελιώδη δικαιώματα που θα διοργανωθεί στο τέλος της χρονιάς. Σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής μας. εγκρίθηκε η άποψη, ε, η πρόταση της ε, Προέδρου. Επίσης, οι συντονιστές ανέθεσαν στην Πρόεδρο να αποστείλει επιστολή στη Σουηδική κυβέρνηση σχετικά με την καταγγελία διακριτικής μεταχείρισης εις βάρος ενωσιακών πολιτών που δεν διαθέτουν τον τετραψήφιο προσωπικό αριθμό. και θα συζητηθεί το θέμα έπειτα από πρώτες που θα υποβάλει η Γραμματεία. Για τις προσβαλόμενες συστάσεις, αυτές εγκρίθηκαν με εξαίρεση την ε, αναφορά 434 του 2018 που ε, ε, ε, χαρακτηρίστηκε παραδεκτή και θα δοθεί συνέχεια. Κλείσαμε την 444 του 2018. Οι αναφορές 254, 695, 1198 παραμένουν ανοιχτές και θα δοθεί συνέχεια σε αυτές. Και μετά, διερευνητική επίσκεψη και ακροασει. Οι συντονιστέ αποφάσισαν να μην διοργανωθούν διερευνητικέ επισκέψεις το πρώτο εξάμεινο του 2019 αλλά αποφάσισαν να διοργανωθεί ε, μια ακρόαση για την κλιματική αλλαγή τον Ιανουάριο του 2019 υπό την προϋπόθεση ότι θα συμμετάσχουν σε αυτή την ε, ακρόαση και καθήλυνα αρμόδιες ε, επιτροπές, η ΕΝΒΙ και η ΙΤΡΕ, κατά προτίμηση και οι δύο, ή τουλάχιστον μία. Επίσης, σχετικά με τη σύνθεση της αποστολής στην Ισπανία αποφασίστηκε η Μπεατρίς Μπεσέρα να είναι η επικεφαλής. Έτοιμα πρασίνων. Για μεταφορά προφορικού ερωτήματος για παραβιάσει του Natura 2000, οι συντονιστέ αποφάσισαν να υποβληθεί προφορικό ερώτημα χωρίς ψήφισμα υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνει σε συνεργασία με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Προετοιμασίε για τη συνάντηση με, τις, ε, ε, με τα Εθνικά Κοινοβούλιο, οι συντονιστές έλαβαν γνώση του επικαιροποιημένου προγράμματος. Και ΦΑΤΚΑ. Οι συντονιστές αποφάσισαν να αποστείλουν ε, επιστολή στην Γερουσία των ΗΠΑ για το ΦΑΤΚΑ και διερευνητική επίσκεψη στον Τιουνιάν. Οι συντονιστές ε, αποφάσισαν να αποστείλουν ευχαριστήρια επιστολή σε εκείνους που δεν καταφέραμε να συναντήσουμε και ε, να τους διαβεβαίσουμε ότι θα λάβουμε υπόψη μας τις γραπτές συνεισφορές που υπέβαλαν. Αυτά όσον αφορά τις αποφάσεις των συντονιστών. Κυρία Μπεσερά, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Muchas gracias. Gracias, presidente. Ευχαριστώ. Και Πρόεδρε, σε σχέση με όσα είπατε για την συνεδρία των συντονιστών εχθές, όπως γνωρίζετε δεν ήμουν παρούσα. Χαίρομαι πάρα πολύ για την απόφασή σας σχετικά με την αποστολή του Δεκεμβρίου θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική για φέτος. Σε σχέση με μία από τις αποφάσεις που λάβατε χθες όμως θα ήθελα να ρωτήσω ή τουλάχιστον να σας προσκαλέσω να σκεφτούμε το εξής. Εχθές μία αναφορά απορρίφθηκε. Η αναφορά σε σχέση με το πώς λειτουργεί η περιφερειακή τηλεόραση και πώς επηρεάζει τους πολίτες. Αναφέρομαι στην, στο κανάλι 3 της καταλανικής τηλεόρασης. Ε, είναι παρόμοια με άλλες αναφορές που έχουν απορριφθεί σε σχέση με έλλειψη ουδετερότητας και σε άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς. Επιτρέπουμε όμως σε άλλους να, να δώσουν το παρόν και να παρουσιάσουν τις αναφορές τους θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι που ε, δεν εξυπηρετεί τα δικαιώματα των πολιτών. Εχθές, παρά το ότι είχαμε συμφωνήσει να ακούσουμε αρχικά την αναφορά αυτή, τελικώς την απορρίψαμε. Ίσως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε σε σχέση με τις αρμοδιότητες αυτής εδώ της Επιτροπής το επιχείρημα ήταν ότι πρόκειται για μια αναφορά πολιτικής χρειάς. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο έχει πολιτική χρειά το γεγονός ότι υπάρχουν παράπονα από πολίτες σχετικά με τη μη ορθή χρήση ενός ε, δημόσιου μέσου. Θα ήθελα να σας προσκαλέσω να προσπαθήσουμε να το σκεφτούμε στα πλαίσια της Επιτροπής μας αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ό,τι αφορά το πρώτο κομμάτι. Σας συγχαίρω για την αποστολή σε ό,τι αφορά το δεύτερο κομμάτι. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο τώρα. Συμφωνήθηκε από τους συντονιστές και δεν έχω κανένα δικαίωμα να παρέμβω στην απόφασή τους. Αντιθέτως, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να σκεφτούμε, γιατί η Ολομέλεια μπορεί να απορρίψει την ε, απόφαση των συντονιστών. Γι' αυτό πιστεύω το ερώτημα αυτό έχει ουσία. Υπάρχουν δύο διαφορετικές αναφορές. Αυτή έχει καταχωρηθεί και πρωτοκολληθεί τον Απρίλιο και λέει ότι δεν υπάρχει διαφάνεια και ότι εκεί υπάρχει, υπάρχουν αναλυθείς συγκεκριμένες πληροφορίες και αναφέρει την Καταλωνία. Μετά είχαμε την άλλη το Σεπτέμβριο τα είπαμε οι συντονιστές και είπαμε να την ε, κάνουμε δεκτή και μόλις ξεκαθαριστεί ότι είναι δεκτή, γιατί είναι θέμα καταπάτης δικαιωμάτων, έχουμε κάποια προηγούμενα τέτοια και ε, αυτό με το συνεργείο της τηλεόρασης. Και όπως είπε και ο Πρόεδρος, πρόκειτο το, για το θέμα του πώς θα φτιάξουμε σε διάταξη, όχι για το θέμα του αποδεκτού. Είπαμε να μην τη βάλουμε και οπότε αυτοί οι δύο αναφέροντες ακούσαν από εμά ότι ναι, παραδεκτή, θα τη μελετήσουμε και όταν είπαμε να τη βάλουμε στην μέση διάταξη ελέγχθη όχι αναβάλλεται παόριστον. Ε, δεν έχει νόημα αυτό, δεν δείχνουμε συνέπεια έτσι. Γι' αυτό και σας ζητάω. Σας ζητάω τώρα να αλλάξουμε απόφαση. Δεν, ξέρω, δεν ξέρω ποιος θα με καλύψει γι' αυτό. Δεν, δεν έχει νόημα αυτό που κάναμε. Ναι, η ολομέλειά μας ούτως υπήρ μπορεί να πει όχι. Όντως. Και κάτι άλλο τώρα. Και κάπου να κάνουν και άλλη αναφορά μετά να επανέλθουν. Επίσης, όσον αφορά τα εγκλήματα της ε, ΕΤΑ, είχαμε αναλάβει δράση και είχαν επίσης συντονιστέ εκτός από το Λαϊκό Κόμμα, όχι. Αυτό να θυμίσω, τίποτα άλλο. Βλέπω, ακούω, σημειώνω την άποψή σας, αλλά εγώ είμαι πρόεδρος και σας επαναλαμβάνω. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να το ξανασυζητήσουμε. Αποφασίστηκε από τους συντονιστές, έχετε δικαίωμα να το ξαναθέσετε το θέμα τον Νοέμβριο, αλλά όχι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ξεκινάμε με τις ψηφοφορίες. Μεταφορά ζώων την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά. Ε, είστε έτοιμοι να περάσουμε στην πληροφορία. Πάμε. Λοιπόν, τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Α, αποχές, με συγχωρείτε. Να το ελέγξουμε σας παρακαλώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. The vote is closed. Πέρας της ψηφοφορίας. Γιατί ψηφίζουμε επί της 6. Ξανά. Ξανα, ξα, ξαναψηφίζουμε επί της 6. Παρακαλώ ψηφίστε. Close the vote. ψηφοφορίας. Και το αποτέλεσμα είναι... Εγκρίνεται. Ό,τι εγκρίνεται. 13 υπέρ 10 κατά. Ε, τροπολογία 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αποχές. Ναι. Τροπολογία 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία της κυρίας Βαλίνα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ, Τροπολογία 4. Ξαναλέω. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λοιπόν συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Yeah. Oral amendment of Madam Valina in favor. Προφορική τροπολογία της κυρίας Βαλίνα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Amendment 20. Τροπολογία 25 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Όχι, να ελέγξουμε, φωνάζουν. Ελέγχουμε, ελέγχουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 25. Ψηφίστε παρακαλώ επί της τροπολογίας 25. And now, close. Πέρας. Απορρίπτεται. 26. Υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Ελέγχουμε. Ψηφίζουμε επί της τροπολογίας 26 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 19 ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 20 δεύτερο τμήμα υπέρ η 26 εγκρίθηκε λοιπόν ξαναπάμε τροπολογία 20 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Όχι. Με συγχωρείτε. Τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Επί της τροπολογίας 42. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της Εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Ναι, παρακαλώ, πείτε μας. Ähm, κύριε Πρόεδρε, ε, στην 21 το δεύτερο τμήμα είναι ε, συμβατό με την 25. Αν ακούσαμε καλά, γιατί ο μιλητής μιλάει πολύ μακριά από το μικρόφωνο. What is it? So, if 25 or 26, one of them is adopted, then this, this, this, and this fall. Yeah. And in the second, in the second part says explicitly. Το δεύτερο τμήμα λέει ο, ε, ρητός ότι είναι συμβατό με τις τροπολογίες 25 και 26. Γι' αυτό και πρέπει να ψηφίσουμε. Μα ψηφίσαμε. Δεν ψηφίσαμε επί του δεύτερου τμήματος. Ψηφίσαμε, λέει ο πρόεδρο. Επαναλαμβάνει ο πρόεδρο. Ψηφίσαμε την τροπολογία 20, το δεύτερο τμήμα. Έγινε ψηφοφορία.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 second parts of the 20 and 21 are identical. Yeah. Thank you. So, we... uh... Ωραία. Το λύσαμε. Συμβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα προφορική τροπολογία. Πάμε της κυρίας Βαλίνα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 12. Υπέρ. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 47. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος, ωραία. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά λοιπόν επί τη τροπολογία 32. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 33. Μόνο το πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική προφορική τροπολογία της Βυρζινή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά Συμβαστική τρία, ξαναλέω. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε στην 37. Τροπολογία 37. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Όχι, εντάξει, απορρίπτεται. 39. 38, συγγνώμη. 38, 38. Υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 39, υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 40, υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 πίπτη. οπότε περνάμε στην τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά επί του συνόλου του σχεδίου γνωμοδότησης πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε τώρα με την έκθεση για τη διερευνητική επίσκεψη στη Λουσατία, στη Γερμανία. Είστε έτοιμοι? Auken. Κυρία Άουκεν, θέλω να σας πω ότι φυσικά θέλω να ε, ψηφίσετε υπέρ της έκθεσης, αλλά ειδικά στην αρχή μιλάμε για το λιγνίτι και θυμηθείτε τι έγινε χθες, όταν λάβαμε αυτήν την δραματική έκθεση του IPCC, που λένε ότι αν συνεχίσετε με την ε, παραγωγή άνθρακα και λιγνίτη, ε, αυτό θα είναι ε, καταστροφή. Έχουμε να κάνουμε με μια κοινωνική καταστροφή που μας περιμένει, αν δεν αναλάβουμε δράση. Θυμηθείτε το αυτό λοιπόν στην ε, στάση σας ε, στις ψηφοφορίες για το περιβάλλον, για το κλίμα. Πρέπει να αναλάβουμε δράση επιγόντως. Κάποιοι από εσά βέβαια δεν πιστεύετε στην κλιματική αλλαγή, δεν πρόκειται να σας πείσω τώρα προφανώς. Μπορείτε να πιστεύετε και στον, ε, και στον Άι Βασίλη άμα θέλετε, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε ευθύνη. Κύριε Πρόεδρε, εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί αναπληρωματικοί. Έχουμε και άλλες ψηφοφορίε να κάνουμε. Μην, μην περνάμε τώρα σε διάλογο και συζήτηση, γιατί έχουμε πολλές ψηφοφορίε και πάρα πολλά θέματα να εξετάσουμε. Ωραία, εντάξει, ψηφοφορία. Πάμε. Διερευνητική επίσκεψη στην Λουσα, Λουσατία. Συμβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, Τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1 υπέρ, εναντίον, αποχές. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, νομίζω ότι δεν εγκρίνεται, άρχεται η ψηφοφορία. Τελείωσε, ολοκληρώθηκε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Εναντίον. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά αποχές. Ελέγχουμε για την τροπολογία νέα ηλεκτρονικά. Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται η τροπολογία νέα. Απορρίπτεται η τροπολογία 9.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 21. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά, λέει ο πρόεδρος, την τροπολογία 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Ολοκληρώνεται. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22. Πρώτο κομμάτι ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Το δεύτερο μέρος της τροπολογίας 22, ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. Ολοκληρώθηκε. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την, ψηφολογία, για την τροπολογία, με συγχωρείτε, 23. Απορρίπτεται. Τώρα, τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική, Ολοκληρώθηκε. Εγκρίνεται με 19 ψήφους. Ευχαριστώ. Θες να κάνω εγώ, Yeah, I, okay, okay, okay, And third, third of our voting is, is concerning ψηφοφορία αφορά τον Ιούγεν. Χαν, τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ελέγξουμε, λέει ο πρόεδρος. Τροπολογία 1, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Απορρίπτεται η τροπολογία 9. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται η τροπολογία 10. Τροπολογία 11. Ξεκινάμε με το πρώτο μέρος, ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, έγκρινεται. Το δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Το πρώτο μέρος ψηφίζουμε υπέρ, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, εγκρίνεται. Με συγχωρείτε. Όχι να... Ψηφίζουμε για το δεύτερο μέρος της τροπολογίας 12. Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία ηλεκτρονική, εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για την τροπολογία η τροπολογία 13 εγκρίνεται λέει ο πρόεδρος να ελέγξουμε την τροπολογία 13 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά Τροπολογία 13. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ολοκληρώνεται την ψηφοφορία. Απορρίπτεται η τροπολογία 13. Τροπολογία 14. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Τροπολογία 15, δεύτερο μέρος. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16, πρώτο μέρος. Υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 16, πρώτο μέρος. Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Το δεύτερο μέρος της τροπολογίας 16. Τροπολογία 16 δεύτερο μέρος. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε και ηλεκτρονικά. Τροπολογία 16 δεύτερο μέρος. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος, τροπολογία 17 δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Τροπολογία 18, υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Τροπολογία 7, υπέρ, με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος. Τροπολογία 19. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές. Κατά πώς φαίνεται απορρίπτεται. Τροπολογία 19 να το ελέγξουμε όλα ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται η τροπολογία. Τροπολογία 20 τώρα. Υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να το ελέγξουμε και ηλεκτρονικά τροπολογία 25 ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία Η τροπολογία 25 εγκρίνεται. Τροπολογία 26 παρακαλώ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 31 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 33 το πρώτο μέρος ψηφίζουμε. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 34 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά, ψηφίζουμε, ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 35. Υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Εγκρίνεται. 37. Εγκρίνεται και 37. 38. Εγκρίνεται. 39. Απορρίπτεται 39. Να το ελέγξουμε. Όχι, προχωράμε. Τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Τροπολογία 40 ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41. Το πρώτο μέρος ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 42 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά τροπολογία 43 ψηφίζουμε ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία εγκρίνεται Τροπολογία 44. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 45. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46. Το πρώτο μέρος. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 47 τροπολογία και 48 είναι πανομοιότυπες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 κατά υπέρ κατά με συγχωρείτε 51 τροπολογία εγκρίνεται. Να την ελέγξουμε και ηλεκτρονικά, την ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 52. Απορρίπτεται. Τροπολογία 53. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 54. Εγκρίνεται. 55. Το πρώτο μέρος ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ, Εγκρίνεται. 56 υπέρ. Με συγχωρείτε τη 57. Το πρώτο μέρος της 57 ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος της τροπολογίας 57 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 59, 60, εγκρίνεται, 61, Απορρίπτεται η 61. 62. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 63. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται την 63 να την ελέγξουμε και ηλεκτρονικά ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία εγκρίνεται και τώρα τελική ψηφοφορία άρχεται η ηλεκτρονική ολοκληρώθηκε εγκρίνεται με 12 ψήφους. Σας ευχαριστώ πολύ.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 Ας προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το της ονομοδότησης που προβλέπεται στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Αφορά τις ε, διατάξεις που ορίζουν τα της λειτουργίας, του λειτουργήματος μάλλον του διαμεσολαβητή. Κύριε Άουκη. Όπως λέγαμε. Τα έχουμε πει τέσσερις φορές στην ε, Ολομέλεια. Θέλουμε να αναθεωρηθεί το καθεστώς που δίνει τον Διομεσολαβητή. Τα λέμε και τα ξαναλέμε. Δεν είναι τα πράγματα όσο στεγνά θα θέλαμε. Και τα βασικά μου θέματα είναι τα εξής. Χρειαζόμαστε διαμεσολαβητή πιο ισχυρό. Οι τρεις που πέρασαν από εδώ ήταν μάλλον εξαιρετικοί, αλλά δεν έχουν αρκετούς πόρους, δεν έχουν αρκετά ισχυρές αρμοδιότητες, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες του κόσμου. Θα σας πω και άλλα δύο-τρία λόγια που μου φάνηκαν αυτά από τα οποία διάβασα σημαντικά. Δηλαδή ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η σωστή διοίκηση. Θα πρέπει να καταπολεμηθούν οι συγκρούσεις συμφερόντων στην διοίκηση. Είναι θέμα ηθικής, αλλά αν κανείς παίρνει αποφάσεις για τον κόσμο, δεν θα πρέπει να υπάρχουν σύγκρουση συμφέροντων. Δεν αρκεί το να δηλώνει κανείς τη σύγκρουση συμφέροντων. Και αυτό είναι πρόβλημα που ανακύπτει συνέχεια. Ε, γι' αυτό και είναι τόσο σημαντικό να δώσουμε τα μέσα στο διαμεσολαβητή. Αλλιώς δεν λειτουργεί ο θεσμός. είναι το δημογόμενο συμφέρονται προς τους ε, περιβαλλοντικούς φορείς, ε, τα αντίθετα συμφέροντα. Ε, θα πρέπει αυτά να ρυθμιστούν, να υπάρχει πρόσβαση ξεκάθαρη στα δεδομένα και θα πρέπει επομένως να προβλέπονται πιο σημαντικές αρμοδιότητες στο καθεστώς που διέπει και θα πρέπει και η Μεσολαβήτρια που απευθύνθηκε ήδη σε εμάς τώρα να καλυφθεί σε κάθε έκθεση που υποβάλλει να ανταποκριθούμε όπως έκανε τώρα για το ότι δεν υπάρχει διαφάνεια στο Συμβούλιο Ξέρετε, Συρλανδία, Σκανδιναβία, Ηνωμένο Βασίλειο, κάτω χώρε υπάρχουν μεσολαβήτε, αλλά άλλο είναι πολύ αδυνατό ε, ο θεσμό. Α πούμε στη Γερμανία ε, υπάρχουν περιφερειακοί. Ε, αλλού επίση δεν είναι ισχυρή σε άλλα κράτη. Οπότε ε, δεν τον βλέπουν και πολύ σοβαρά λένε, α, σαν να είναι πρόεδρος μιας επιτροπής να εντοπίζουν. Δεν είναι έτσι όμως. Είναι κάτι διαφορετικό, θα πρέπει να είναι αυτός ανεξάρτητος. Είναι σαν δικαστής. Θα πρέπει όλα αυτά να αναδειχθούν πιο ξεκάθαρα από όσο τώρα. Και ο κόσμος να ξέρει, να εμπιστεύεται το θεσμό. Ότι έχει κάποιον δηλαδή να του προστατεύει τα συμφέροντα. Επίσης, είναι περίεργο. Να μπορεί, να μπορεί, να μπορεί να πάρει και σε δικαστήριο. Οπότε θα πρέπει τώρα να συνειδητοποιήσουμε ότι πρόκειται για ζήτημα σοβαρό. Δεν κατακλείδη. Σας τονίζω ότι επίσης συζητούμε για τους καταγγέλλοντες σε κάθε επίπεδο. Καμιά φορά όμως δεν μπορεί να γίνει η διάκριση αν κάποιος καταγγέλει κάτι ή αν προσφέρει απλώς και ζητάει συμβουλή ε, για να οργανώσει τη δουλειά του ή... Α, να υπάρχει κατάλληλη προστασία. Ε, στα λόγια ωραία τα λέμε. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει περιβάλλον σίγουρο. και διαμεσολαβητής δεν είναι τίτλος, είναι λειτουργήμα. Ξέρετε, και αυτή η λέξη ombudsman είναι, έχει ρίζες ιστορικές στη Σκανδιναβία, στη γλώσσα. Αυτό είναι το βασικό που ήθελα να αναδείξω στο κείμενό μου. Και βέβαια Όποιος θέλει μπορεί να συμβάλλει να βελτιώσουμε το κείμενο. Ο Πρόεδρος. Να δώσουμε τώρα το λόγο στους κοιόδης συγητές. Βίλαντ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Άουκεν για το σχέδιο γνωμοδότησης. Είναι πραγματικά πολύ σωστό μετά από τόσα χρόνια να εξετάσουμε μια αναθεώρηση της νομικής βάσης επί της οποίας ε, ενεργεί και δραστηριοποιείται ο διαμεσολαβητής. Πιστεύω και εγώ ότι ο διαμεσολαβητής πρέπει να έχει μεγαλύτερη πρόσβαση σε έγγραφα προκειμένου να μπορεί να σχηματίζει εικόνα για τις υποθέσεις που επεξεργάζεται. Ωστόσο, δεν ξέρω αν ήταν πρόβλημα της διερμηνίας, ε, αλλά ε, ακούστηκε ο όρος δικαστής. Εγώ πιστεύω ότι σε ό,τι και αν κάνουμε πρέπει να γίνονται σεβαστές οι αρχές της διάκρισης των εξουσιών. Οι αρχές διάκρισης των εξουσιών έχουν αποδειχθεί ως πολύ αποτελεσματικέ και ο διαμεσολαβητής ή η διαμεσολαβήτρια δεν είναι ουδέτερη αρχή. Σκοπός του διαμεσολαβητή είναι να βοηθά τους πολίτες. Στην υπηρεσία των πολιτών λοιπόν και γι' αυτό θα πρέπει να είναι και αμερόληπτος. Η εντύπωση που αποκόμισα από τα όσα μας είπε η κυρία Άουκεν είναι ότι ο διαμεσολαβητής θα είναι ε, μια πόλα. Αστυνομικός, ε, δικαστής, ε, ενδεχομένως και πληρεξούσιος ε, των δικαστηρίων για την εκτέλεση αποφάσεων, να μπορεί να κάνει τα πάντα και βεβαίως να κυνηγάει τους κακούς αυτού του κόσμου. Ε, αυτό νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολική προσέγγιση. σε σχέση με τον ρόλο που πρέπει να αποδοθεί στο διαμεσολαβητή και είναι και λίγο υπερβολική προσέγγιση αυτή ως προς το τι μπορεί να επιτύχει ένας δημοσιογραφητής. Αναφέρθηκε η συγκήτρια και στο, θέμα των πληροφοριοδοτών, των κατεγγελόντων. whistleblower. Ένας πολίτης που ε, θεωρεί ότι μπορεί να είναι πληροφοριοδότης, μπορεί και να μην έχει πολύ ξεκάθαρη εικόνα για το τι κάνει. Τι γίνεται όμως όταν έχουμε έναν πληροφοριοδότη ο οποίος εργάζεται σε έναν οργανισμό ο οποίο δεν είναι καταχωρημένο στο Μητρό Διαφάνειας. Ποιο θα τον υποδεχθεί αυτόν τον άνθρωπο αν υπάρχουν τόσο σημαντικές και τόσο αυστηροί κανόνε για τη διαφάνεια. Μπορεί να πάει ούτε στην Κομισιόν, ούτε να πάει στην, ε, σε κάποιον Ευρωβουλευτή να απευθυνθεί, γιατί δεν θα είναι καταχωρημένη η εταιρεία του. Κατά τη γνώμη μου αυτό σημαίνει ότι ούτε με το διαμεσολαβητή ένα τέτοιο άνθρωπος έχει τη δικαίωμα να συναντηθεί. Ίσως ε, θα πρέπει και αυτό να το δούμε. Εν πάση περιπτώσει, οι ειδικέ μου τροπολογίε θα επικεντρώνονται στο να υπάρξει βελτίωση των όρων εργασία του διαμεσολαβητή ε, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη αρχές ε, όπως είναι η διάκριση των εξουσιών που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται σεβαστές. Thanks um, um, Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να σας πω από πλευράς της ε, Βιρζινή ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Καλά έπρεπε να φύγει γιατί πρέπει να προεδρεύσει ε, μία συνάντηση για την Γιούριο Σόφρα, την προστασία των ε, ε, καταγγελόντων. Όπως βλέπετε εδώ πέρα επικαλύπτονται τα θέματα. Οπότε πρέπει να ευχαριστήσουμε την Μάργκριτ. Είναι πάρα πάρα πολύ σωστό το κείμενό της όσον αφορά ε, τη δύο μεσολαβήτρια. Οπότε θα πρέπει ε, να σας πω ότι είμαστε δύο μήκος κύματος. Ε, έτσι δεν θέλουμε να υπάρχει σωστή διοίκηση, χρηστή, με διαφάνεια και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα από τις κοινέ μάχες που έχουμε δώσει για αυτές τις ε, βασικές αξίες. Έχουν πέρασει 10 χρόνια από την τελευταία φορά που τροποποιήθηκε το καθεστώς που διέπει τον διαμεσολαβητή. Πολλά έχουν γίνει. Οπότε νομίζω ότι όντως ε, είναι βάσιμη η πρόταση της ε, Μαργαρίτ. πολύ σωστές οι ιδέες της σε σχέση με το πώς θα πρέπει να αλλάξει το τι ισχύει. Ναι, ε, την υποστηρίζουμε για τα έγγραφα, για τη διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας. Τώρα και διαφοροποιούμαστε όσον αφορά την πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και για τα έγγραφα ε, συμφωνούμε για, με την ομολογία του δικαστήριου και με τον κανονισμό του 2001. Ε, επίσης θα πρέπει να δούμε τι ισχύει με τη σεξουαλική παρενόχληση στα θεσμικά όργανα, τι μπορεί να κάνει ο διαμεσολαβητής, να δούμε πώς θα αναβαθμιστεί η συνεργασία μας με τον διαμεσολαβητή ε, και βεβαίως το να μπορεί να προσέρχεται και να συμμετέχει στην ε, Ολομέλεια. Επίσης το ίδιο ισχύει, δηλαδή συμφωνούμε με την προστασία των καταγγελόντων και βέβαια θεωρούμε ότι και εδώ μπορούμε να τροποποιήσουμε τις κείμενες διατάξεις. Μπράβο λοιπόν στην εισηγήτρια, θα συνεργαστούμε μαζί της και με τους άλλους συνάδελφους και όδους εισηγητής για το θέμα. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Μαριά. Κύριε Πρόεδρε, Θεωρώ ενδιαφέρουσα την έκθεση και το γεγονός ότι συζητούμε για το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Να πω ότι το 1993 όταν ξεκίνησε όλη η διαδικασία με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή είχα την ευκαιρία να γράψω το πρώτο βιβλίο που έχει γραφεί για την έννοια και το ρόλο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και να κάνουμε και ένα συνέδριο στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης του Μάστριχτο που ήμουν senior lecturer. Από τότε πέρασαν χρόνια βεβαίως και νομίζω ότι η εμπειρία που έχει σωρευτεί μας δίνει τις εξής σκέψεις για να πάμε παρακάτω. Πρώτα απ' όλα ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι. Γιατί σε διάφορες ε, γλώσσες σημαίνει κάτι διαφορετικό. Διαμεσολαβητής ε, στα ελληνικά σημαίνει μεσολαβό ανάμεσα σε δύο αντικρουόμενα συμφέροντα. Όμως η έννοια του διαμεσολαβητή, δηλαδή του ombudsman, έχει άλλο χαρακτηριστικό καθώς προέρχεται από τη Σκανδιναβία. Είναι ένα είδους ε, defensor del pueblo θα έλεγε κανείς στα ισπανικά, δηλαδή είναι αυτός που στηρίζει τον πολίτη απέναντι στην ισχυρή διοίκηση και στα φαινόμενα κακοδιοίκησης. Γι' αυτό χρειάζεται μια πολιτική στήριξη και η πολιτική στήριξη του ομπουτσμάν του διαμεσολαβητή γίνεται από το Κοινοβούλιο. Γίνεται εν προκειμένου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό και διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολιτικά να στηρίζει τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή στη σύγκρουση που θα κάνει με τα όργανα της Ένωσης για να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα κακοδιοίκησης. Άρα ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής βεβαίως θα είναι ανεξάρτητος, θα είναι αμερόληπτος, αλλά πρέπει πολιτικά να στηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην έννοια της κακοδιοίκησης πρέπει να δούμε τι σημαίνει κακοδιοίκηση και ποιες είναι οι δράσεις που πρέπει να ελέγξει. Φερρυπίν, η σύγκρουση συμφερόντων, καθώς ανακύπτει σήμερα, είναι κλασική μορφή κακοδιοίκησης. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και σε επίπεδο κομισιών και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εν προκειμένου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει σύγκρουση συμφερόντων κατά την άποψή μου που συμμετείχε και ως μέλος της Τρόικας και έπρεπε να ενεργεί με βάση τις εντολές του Eurogroup αλλά ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητη αρχή και άρα πρέπει να μην δέχεται εντολές. Άρα δεν μπορούσε να ενεργεί ως Τρόικα που δεχόταν εντολές από το Eurogroup. Αυτό λοιπόν είναι ένα σοβαρό ζήτημα σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό λοιπόν το θέμα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Το δεύτερο είναι η διαφάνεια και η λειτουργία των οργάνων. Σήμερα το πιο ισχυρό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το Eurogroup. Αυτό παίρνει τις πιο σημαντικές αποφάσεις. Αυτό επηρεάζει τη ζωή την καθημερινή των πολιτών. Και όμως ουσιαστικά το Eurogroup είναι ανεξέλεγκτο. Κάποιο πρέπει να ελέγξει τι δραστηριότητέ του. Και αυτό οπωσδήποτε πρέπει να είναι ο ίδιο ο διαμεσολαβητή αλλά ο διαμεσολαβητής πρέπει να ελέγξει και την κακοδιοίκηση εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Yes, I, I will listen to your comments later, but listen to my comments also. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής πρέπει να ελέγξει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να σας φέρω ένα παράδειγμα κύριε Αντιπρόεδρε. Υπάρχει μια διαδικασία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν υποβάλλουμε ερωτήσεις οι οποίες ελέγχονται από το επίπεδο του Προέδρου αν αυτές είναι εντός λέει της αρμοδιότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πολλές ερωτήσεις μας επιστρέφονται για να τις ξαναγράψουμε. Εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι μορφή κακοδιοίκησης και θα μπορούσε να ελεγχθεί αυτή η μορφή κακοδιοίκηση από τον ίδιο τον Ombudsman. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει ο διαμεσολαβητής θεωρώ σημαντικό το γεγονός να μπορεί να παρίσταται ο διαμεσολαβητής και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν το ζητήσει και στις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν το ζητήσει αλλά να μπορεί να έχει και δικαίωμα παρέμβασης εντός του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή να παρεμβαίνει σε υποθέσεις που θεωρεί ότι πρέπει να υποστηριχθούν και κατά την άποψή μου αυτό το δικαίωμα πρέπει να το πάρει. Ένα άλλο θέμα είναι η πρόσβαση στα έγγραφα, που νομίζω ότι είναι σοβαρό. Ένα άλλο ζήτημα είναι η προστασία των καταγγελόντων, κάτι το καινούριο, το διαφορετικό σε αυτή τη φάση. Όπως βεβαίως και το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης, το οποίο έχει, αν θέλετε, έρθει πλέον στο προσκήνιο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ο προβληματισμός είναι διάχυτος. Βεβαίως μέσα από τις τροπολογίες και τις δικές μας και των υπολείπων θα κάνουμε ένα διάλογο επί της ουσίας του τι θέλουμε να ισχύσει και από εκεί και πέρα βεβαίως θεωρώ ότι σε βασικές γραμμές η έκθεση της κυρίας Άουκεν πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα και εμείς θα κάνουμε τις δικές μας τροπολογίες. Ευχαριστώ. Πασκάλ Λεφέμπρ Πασκάλ Λεφέμπρ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι, ευχαριστώ. Καταρχάς θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Όκεν για το έργο που έχει επιτελέσει σε αυτό το θέμα. Ορθώς επισημαίνεται ότι το Κοινοβούλιο έχει πολλάκι ζητήσει την αναθεώρηση του καθεστώτος και είναι επίσης αλήθεια ότι ε, μερικές φορές τα πράγματα έγιναν με το κεφάλι ανάποδα. Γιατί ξέρετε ότι ε, έγινε αναθεώρηση του, της εκτελεστικής απόφασης του 2016. Αντί λοιπόν να αναθεωρηθεί η πρώτα το καθεστώς και στη συνέχεια οι εκτελεστικές διατάξεις, έγινε ανάποδα. Ίσως από άποψη μεθοδολογία δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή λύση. Ξέρετε ότι οι σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι εξαιρετικέ και φυσικά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Διαμεσολαβητής καθώς και άλλα θεσμικά όργανα και φορείς ε, αποτελούν ένα αντίβαρο ε, στην άσκηση των εξουσιών και αυτό είναι πολύ θετικό συνολικά για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Γνωρίζουμε ότι η Κομισιόν θα πρέπει να υποβάλει τη δική της γνώμη βεβαίως για το θέμα αυτό. Το 2019 θα γίνει αυτό, αν ε, καταφέρουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα και αυτό θα είναι μια ευκαιρία να εξετάσουμε ε, σε βάθος όλες τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί σχετικά με την αναθεώρηση του καθεστώτος του διαμεσολαβητή. Ωστόσο, Μπορώ να κάνω κάποιες ε, προκαταρκτικές παρατηρήσεις, μη δεσμευτικού χαρακτήρα όμως. Όσον αφορά τις τροπολογίες ε, της Επιτροπής σας. Όσον αφορά την έδρα του διαμεσολαβητή ε, εδώ στις Βρυξέλλες, να σας πω χωρίς να λαμβάνουμε κάποια συγκεκριμένη θέση, να σας υπενθυμίσω ότι η κυρία Οράιλι, ήδη ε, περνά τον περισσότερο καιρό της στις ε, Βρυξέλλες και τα δύο τρίτα των ε, υπαλλήλων που επεξεργάζονται τις υποθέσεις που λαμβάνει ο διαμεσολαβητή εργάζονται στη Ρήμοντο του εδώ δίπλα στι Βρυξέλλες. Επίσης, όσον αφορά το, το δικαστήριο, πάλι μια προκαταρκτική παρατήρηση να κάνω. Έχουμε κάποιες αμφιβολίες όσον αφορά τι τροπολογίε και τι προτάσει που έχουν υποβάλει κάποιοι ευρωβουλευτέ τη Επιτροπή Αναφορών, διότι πιστεύουμε ότι ο διαμεσολαβητή έχει πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Και μ' αρέσει ο όρο στα γαλλικά που είναι ο ε, όρο mediateur. Θα πρέπει λοιπόν να το σκεφτούμε διπλά. Προτού δώσουμε τη δυνατότητα στο διαμεσολαβητή να, να αναλάβει και έναν άλλο ρόλο πλην της διαμεσολάβησης μεταξύ των θεσμικών οργάνων και της εξέβρεσης λύσεων σε προβλήματα. Ε, προτού δηλαδή προχωρήσουμε και του αναθέσουμε και ένα πιο συγκρουσιακό ρόλο αν θέλετε. Επίσης, υπάρχουν ε, προτάσεις σχετικά με τις συστάσεις για την εφαρμογή των αποφάσεων του δικαστηρίου. Έχουμε την εντύπωση ότι αυτές οι συστάσεις δεν θα τηρούνται πάντοτε, ακόμα και αν ε, του αποδοθεί ένας τέτοιος ρόλος. Βεβαίως, συμπάσχουμε όσον αφορά ε, τις ε, διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση σεξουαλικής παρενόχλησης. Γι' αυτό και περιμένουμε να δούμε τι θα περιλαμβάνει αυτή η διαδικασία fast track που θα προταθεί ε, η οποία θα συμπληρώνει ή θα αντικαθιστά το άρθρο 19 του κανονισμού του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως προσβλέπουμε ε, και περιμένουμε να, να, να παραλάβουμε τη σχετική πρόταση και να την εξετάσουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Όσον αφορά τις προθεσμίες που έχουν τεθεί, Μα λέτε ότι θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένε ε, προθεσμίε όσον αφορά τι ε, τροπολογίε που θα υποβληθούν. Να σα υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώ και όλα τα άλλα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα, υπόκεινται σε πολύ αυστηρότερες προθεσμίες με τους νέους κανόνες. Κάποιες φορές πρέπει να πατήσουμε εντός και ε, λίγων εβδομάδων, εντό ενός μήνα, δύο μηνών, τριών μηνών. αλλά αντιστοίχω δεν υπάρχουν ε, προθεσμίες για το διαμεσολογητή εντός των οποίων θα πρέπει να μας απαντήσει και να έρθει σε μας με γνωμοδότηση. Κάποιες φορές περιμένουμε έναν και δύο χρόνια από τον, ε, για να πάρουμε απάντηση από το διαμεσολαβητή, για να ξέρουμε και τι θα πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια. Ίσως λοιπόν μια καλή ιδέα θα ήταν να ε, επιβάλλονται συγκεκριμένε προθεσμίε και στον διαμεσολαβητή. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο που θα ενισχύσει ή θα βελτιώσει, εν πάση περιπτώσει, τη χρηστή διοίκηση. Τέλος, Βεβαίως είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο ε, εξετάζει στενότερα ε, το τι κάνουν οι υπηρεσίε του διαμεσολαβητή, γιατί πάντα τίθεται αυτό το ερώτημα ποιος θα ελέγξει τον ελεγκτή. Και ποιο θα ελέγξει εκείνον που ελέγχει και ε, διενεργώντας τον, τον έλεγχο. Για παράδειγμα το, το ερώτημα είναι αν συμβεί κάτι στο γραφείο του διαμεσολαβητή και θέλει να υποβάλει ε, μια κακοδιαχείριση σε κάποιον, ε, μια καταγγελία κακοδιαχείρισης ε, για ζητήματα που αφορούν το ίδιο το γραφείο του διαμεσολαβητή. Σε αυτά ακόμα δεν έχουμε απάντηση, δυστυχώς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ να βάλω το λιθαράκι μου για αυτό τον προβληματισμό που είναι πολύ σημαντικός. Και το σχέδιο μένω. Δεν με απασχόλησε προηγουμένω γιατί ασχολιόμουν με τα θέματα των σκιωδών και φυσικά και σύμφωνα με τα όσα είπε η συνάδελφος Σάουκεν πρέπει να αλλάξουν το καθεστώς του διαμεσολαβητή ακριβώς όπως ε, ελεγχθεί. Ναι, με τον λέμε και στα ε, Ιταλικά όμως είναι σωστό το να λέγεται και ε, διαμεσολαβητής να λέγεται επίσης ο υπερασπιστής του πολίτη είναι πιο κοντά στον πολίτη. Οπότε θα πρέπει να αναδείξουν περισσότερο το ρόλο του. Θα πρέπει επίσης να έχει πιο εύκολα πρόσβαση στα έγγραφα της Ένωσης. Οπότε πολύ καλή η προσέγγιση της ε, συναδέλφου. Επίσης ε, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πολλές φορές συμβαίνει το να απορρίπτει η προσφυγή κάποιου στο δικαστήριο της Ένωσης, οπότε θα πρέπει να μπορεί κάτι να κάνει σε αυτή την περίπτωση ο διαμεσολαβητής. Θα πρέπει επίσης να του δώσουμε περισσότερες αρμοδιότητες ε, και για τη σεξουαλική παρενόχληση και για την προστασία των καταγγελόντων. Έτσι, να υπάρχουν οι προϋποθέσεις να μπορεί να παρέμβει ο διαμεσολαβητής όσον αφορά τη διεκπαιρέωση των ε, καθηκόντων τους ε, στους ε, δημόσιους οργανισμούς και θεσμούς. Οι τροπολογίες μας θα έρθουν να αναβαθμίσουν το κείμενο γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικός ο ρόλος του διαμεσολαβητή, ιδίω σήμερα. Θα πρέπει να υπάρχει χαστή διοίκηση σήμερα που είναι σε αυτή τη συγκυρία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να δει ο λαβητής τέλος πάντων, ο υπερασπιστής του πολίτη. Πριν ξαναδώσουμε το λόγο στην κυρία Άουκεν. Θέλει κάποιος άλλο το λόγο. Όχι από ό,τι φαίνεται. το λόγο κυρία Σιγήτρια. Στα Δανέζικα. Ευχαριστώ. Ε, μας λένε οι διερμηνείς ότι καλό είναι να μιλάμε στη μητρική μας γλώσσα, οπότε θα μιλήσω δανέζικα. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους για τα θετικά τους ε, σχόλια. Ο κύριος Βίλαν ήταν εδώ, έφυγε, είχε τι περισσότερε αντιρρήσει. Δεν με εκπλήσει όμω, διότι η Γερμανία δεν ξέρει τι θα πει διαμεσολαβητή. Δεν έχουν διαμεσολαβητή. Υπάρχουν δύο-τρία κρατήδια της Γερμανίας που έχουν ε, κάτι σαν συνήγορο του πολίτη, αλλά δεν έχουν κάτι αντίστοιχο. Και στι τελευταίε εκλογές, ε, μάλιστα, ε, υπήρχαν και υποψήφοι ε, βουλευτέ οι οποίοι ήταν ε, μεσολαβητές. Εμείς είχαμε σοκαριστεί όταν το ακούσαμε αυτό, ότι μπορεί κανείς να είναι στην πολιτική αρένα δηλαδή και ταυτόχρονα να είναι και διαμεσολαβητής και μάλιστα χωρίς να έχει περάσει μια περίοδος ε, μεταβατική, cooling off. Και μάλιστα κάποιος είπε και όλας ε, τότε στις εκλογές ότι ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι ανεξάρτητος όσο και ένας επίτροπος. Τι να πω δηλαδή, τι, τι, να σχολιάσει κανείς. Γεγονός είναι ότι ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι ουδέτερος. Δεν είναι δικαστής, αλλά θα πρέπει να είναι αμερόληπτος και ουδέτερος, αντικειμενικός στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Αυτό πρέπει να το έχουμε να το, και να το διαφυλάσσουμε ως κόρη οφθαλμού, διότι διαφορετικά δεν έχει νόημα να έχει κανείς διαμεσολευτής. Όπως είπε και ο, ε, ε, ο, ο, εκπρόσωπος Κομισιόν, χρησιμοποιείται όρος mediateur στα γαλλικά, διαμεσολαβητής. Αυτό όμως είναι πολύ διαφορετικό, αν θέλετε, ως προσέγγιση από, τον, από την έννοια του Ombudsman. Αυτό που είναι το βασικό καθήκον και υποχρέωση του διαμεσολαβητή είναι να εξασφαλίζει την τήρηση του νόμου και να συνδράμει τους πολίτες όταν εκείνοι καταγγέλουν ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά τους ή η κείμενη νομοθεσία. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο διαμεσολαβητή πρέπει πάντοτε να παίρνει το μέρο του πολίτη όταν θεωρεί ότι δεν έχει δίκαιο ο πολίτη. Γιατί κάποιε φορέ μπορεί να έρθει ένα να καταγγείλει κάτι, μπορεί και να κλαίει ακόμη με δάκρυα στα μάτια, αλλά να διαπιστώσει ο διαμεσολαβητή ότι δυστυχώ δεν έχει δίκαιο ο άνθρωπο αυτό. Διότι αυτό που του συμβαίνει προβλέπεται από την νομοθεσία. Και αυτές τις ικανότητες λοιπόν πρέπει να τις έχει ο διαμεσολαβητής. Αυτό εννοώ με τον όρο αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Μιλούμε λοιπόν για το καθεστώς του διαμεσολαβητή. Εμείς μιλάμε εδώ για την εξασφάλιση της αμεροληψίας, τη αντικειμενικότητα του διαμεσολαβητή. Από κομματικά συμφέροντα, από επιχειρηματικά συμφέροντα για να μπορεί κάθε πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει την αίσθηση και την πεποίθηση ότι θα τύχει τουλάχιστον δίκαιης μεταχείρισης αν προσφύγει στο διαμεσολαβητή. Ε, να σου πω ότι το καθεστώς που διέπει σήμερα τον διαμεσολαβητή καθιερώθηκε πριν από τη Λισαβόνα, τη συνδίκη της Λισαβόνας. Ο 1049. Γι' αυτό και πρέπει να γίνουν αυτές οι, οι αν θέλεις. Και να ληφθούν υπόψη και άλλες εξελίξεις, όπως είναι για παράδειγμα η κατάρτιση του χάρτη θεμελιωδιών δικαιωμάτων. Από αυτή την άποψη πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του διαμεσολαβητή. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να εμένουμε τώρα στον 1049. Λοιπόν, μεροληψία. Αν δεν μπορούμε να ε, μιλήσουμε για θέματα μεροληπτικής μεταχείρισης στο Eurogroup είναι πραγματικά ένα θέμα που πρέπει να το, να το συζητήσουμε και να το εξετάσουμε πάρα πολύ σοβαρά. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής είναι ο μόνος διαμεσολαβητής, νομίζω στην Ευρώπη, που έχει το δικαίωμα να ασκεί κριτική στο Κοινοβούλιο. Κανένας άλλος συνήγορος του πολίτη στην, ε, στην Ευρώπη δεν έχει τέτοιο δικαίωμα. Εγώ ήμουν βουλευτή στη Δανία 25 χρόνια. Είχα πολύ συχνές επαφές με το διαμεσολευτή μας και σας διαβεβαιώ ότι ο διαμεσολευτή της Δανία δεν επιτρέπεται να ασκήσει κριτική στο Κοινοβούλιο της Δανία. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να γίνεται το ίδιο στην Ευρώπη. Καλώ ο Ευρωπαίος διαμεσολευτής έχει το δικαίωμα να ασκήσει κριτική και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θετικό είναι αυτό. Πολλοί μάλιστα ε, είχαν ε, προσβληθεί από τη στάση του Έλληνα συνηγόρου ε, που είχε ασκήσει κριτική εδώ στο Κοινοβούλιο. Κακός, Κακώ είχαν προσβληθεί. Αυτός είναι ο ρόλος του. Είναι λοιπόν ο ρόλος του διαμεσολαβητή να επιτελεί το μεγαλύτερο, τον, τον σημαντικότερο δυνατό ρόλο για τους πολίτες. Και, και σε αυτό το ε, σε αυτόν τον ρόλο του πρέπει να τον συνδράμουμε και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν υπάρχουν συγκρούσει συμφερόντων στο, στην υπηρεσία του δημοσιολαβητή, τότε φυσικά αυτά θα πρέπει να βγαίνουν στο φω. Δεν θα πρέπει να αποκρύπτονται. Αλλά είναι πραγματικά, πρέπει να το πω αυτό, πολύ εμ, ανακουφιστικό να ακούμε τα, την Επιτροπή να ισχυρίζεται ότι δυστυχώς το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε μια κεντρική κυβέρνηση στην Ευρώπη. Ο διαμεσολαβητή όμως έχει προβάδισμα, έχει ηγητική θέση. στην ε, υπεράσπιση της νομοθεσίας. Υψηλότερο ρόλο και από την ίδια την Κομισιόν. Εν περιπτώσει, Όσον αφορά τη μεταφορά τη της ε, έδρα εδώ στι Βρυξέλλε, εντάξει, αυτό συνδέεται και με εξοικονόμηση πόρων. Δεν ε, νομίζω ότι ε, είναι κάτι αρνητικό αυτό. Για την πρόσβαση στα δικαστικά έγγραφα ε, νομίζω ότι είναι ε, επίση πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Δεν είναι δυνατόν διάφοροι οργανισμοί και θεσμικά όργανα να έχουν δικαίωμα πρόσβαση σε δικαστικά έγγραφα και να μην έχει τέτοια πρόσβαση ο διαμεσολαβητή Μου το είπε και ο, Δαν, και ο Δανός διαμεσολαβητής. Είναι απίθανο αυτό τώρα. Ο, μόνος, ο, μόνο, η μόνη υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει πρόσβαση σε δικαστικά έγγραφα είναι ο διαμεσολαβητή. Μα πώ γίνεται αυτό. Αν, αν ένα υπήρχε που θα έπρεπε να έχει πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα, ε, είναι ο διαμεσολαβητή ακριβώς για να μπορεί να εξετάζει σε μεγαλύτερο βάθος τις υποθέσεις που επεξεργάζεται. Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό οπωσδήποτε με την Κομισιόν. Εντάξει, να ακούσω βεβαίως και τις απόψεις που θα μου πούν, αλλά πραγματικά πρέπει να εξασφαλιστεί να, να, να αλλάξει και αυτό το καθεστώς. Επιτέλους να δοθεί πρόσβαση στο διαμεσολαβητή, στα δικαστικά έγγραφα. Ε, και ε, συνολικότερα υπέρ των πολιτών μας φυσικά. Ευχαριστώ. Ε, μου επιτρέπετε συνάδελφοι να σας πω κάποια στοιχεία. Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 11η Οκτωβρίου στις 15 το απόγευμα και η ψηφοφορία θα γίνει στις 21 Νοεμβρίου. Σας ευχαριστώ όλους και κυρίως την κυρία Άουκεν. Λοιπόν, Ευχαριστώ. Και τώρα. Έχουμε μία μελέτη της ε, Επιτροπής μας που την ε, παρήγγειλε. Κρίστιαν Νάγκλ Καλώς ορίσατε, το λόγο. Okay, thanks a lot. Uh, and thanks a lot also to inviting me. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να σας ε, κάνω αυτή την παρουσίαση για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, τις βέλτιστες πρακτικές, πιθανές λύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ και τον Τζόρτζο Μούσα που μας ζήτησε να ε, διεκπαιρεώσουμε αυτή τη μελέτη. Λοιπόν, τα ερώτηματα που προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στη μελέτη μας ήταν πρώτον ε, μια επισκόπηση σχετικά με το νομικό καθιστώς ε, για τον ατμοσφαιρικό αέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι η κατάσταση των διαδικασιών επί παραβάση, γιατί υπάρχουν και κάποιες τέτοιες διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει λόγω της ε, παραβίασης των οριακών τιμών για την ποιότητα του αέρα. Επίσης, εξετάσαμε στενότερα πέντε αναφορές από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, προσπαθήσαμε να αναλύσουμε ποια είναι τα βασικά προβλήματα ε, στην περίπτωση αυτών των αναφορών, αξιολογήσαμε την κατάσταση, ε, κοιτάξαμε τα επίπεδα της ποιότητας του αέρα και επίσης εξετάσαμε και κάποιες βέλτιστες πρακτικές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν ε, τις πόλεις των αναφερόντων, αυτών των συγκεκριμένων των πέντε αναφορών, αλλά και όλες τις πόλεις στην Ευρώπη. Και τέλος, ε, προχωρήσαμε και στην κατάρτιση ορισμένων σύντομων συστάσεων για τις πόλεις που αναλύσαμε. Λοιπόν, νομική κατάσταση είναι η εξή. Υπάρχουν οριακέ τιμέ για ατμοσφαιρικού ρήπου στην οδηγία για τον ατμοσφαιρικό αέρα, την 2008 του 50, καθώ και στην ε, τέταρτη απόφαση πλαίσιο. Υπάρχουν κάποια προβλήματα συμμόρφωσης λόγω υπέρβασης των PM10, οριακών τιμών των, ε, του διοξιδίου του αζότου και σε κάποιες μικρές περιοχές και για, για υπέρβαση των ορίων ε, του διοξιδίου του θείου. Κυρίως όμως έχουμε να κάνουμε με τα σωματίδια 10, τα PM10 και το διοξίδιο του αζότου. Γι' αυτό και η Κομισιόν ξεκίνησε διαδικασία επιπαραβάση ε, εναντίον 16 κρατών μελών για την παραβίαση των οριακών τιμών για τα PM10 και εναντίον 13 κρατών μελών για υπέρβαση των ορίων για το διοξίδιο του αζότου. Πολύ πρόσφατα, νομίζω το Μάιο αν δεν κάνω λάθος, έξι κράτη-μέλη παραπέμφθηκαν στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τρία από αυτά λόγω ε, παραβίασης των ορίων PM10, τρία για, τα, ε, το διοξίδιο του αζότου. Στη Βουλγαρία και στην Πολωνία ήδη έχουν ξεκινήσει τέτοιες διαδικασίες εδώ και αρκετό καιρό και μάλιστα ελήφθηκε απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το οποίο, η οποία αναφέρει ότι οι δύο αυτές χώρες παραβιάζουν την ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Λοιπόν, οι αναφορές που εξετάσαμε εμείς στις μελέτες μας και που μας τις διαβίβασε ο κύριος Μούσα κάλυπταν την Ισπανία, τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια, αυτές τις δύο πόλεις, όπου ήδη από το 2011 χρονολογούνται αυτές οι αναφορές. Εκεί αναφερόταν η αναφορά αυτή στο ότι υπάρχει ε, παραβίαση της οδηγίας 2008 τους 50 από το Δήμο της ε, ε, Μαδρίτης. Υπήρξε, εξετάσαμε και μια αναφορά για την Αμβέρσα, που αφορούσε την Αμβέρσα και εμείς εξετάσαμε και τις Βρυξέλλες. Στην Ιταλία εξετάσαμε την περιοχή της Λομβαρδίας, του Μιλάνου και στη Γαλλία εξετάσαμε μια αναφορά που αφορούσε την Μασαλία και το Παρίσι. Λοιπόν, εξετάσαμε καταρχάς τα προβλήματα της τάσης που παρατηρούνται στις πόλεις όσον αφορά τα επίπεδα της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Υπάρχουν, ε, πολλά, ε, υπάρχουν ε, πολλές θετικές εξελίξεις σε πολλές πόλεις, βελτιώνεται η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ωστόσο εξακολουθούμε να διαπιστώνουμε υπερβάσεις για τα PM10 στη Λομβαρδία για παράδειγμα υπάρχουν πάρα πολλές μέρες κατά τη διάρκεια ενός χρόνου όπου εμφανίζονται υπερβάσεις αν και το ετήσιο όριο η Λομβαρδία το τηρεί, το ετήσιο. Στις μεγάλες πόλεις, στα μεγάλα αστικά κέντρα φαίνεται ότι εξακολουθούμε να, υπάρχουν, να, να αντιμετωπίζουμε κάποιες μέρες όπου ε, υπάρχουν σημαντικές ε, υπερβάσεις των PM10. Το ίδιο και στη Βαλένσια. Στην, στο στο, στην περίπτωση του διοξιδίου του αζότου δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι τόσο θετικά όσο ε, ε, στην περίπτωση των σωματιδίων. Όλες, με εξαίρεση τη Βαλένθια, υπερβαίνουν σημαντικότατα τις οριακές τιμές. Η τάση είναι πτωτική, αλλά ή στάσιμη, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της, ε, της Μαδρίτης και της Μασαλίας. Στάσιμη ή πτωτική παρόλα αυτά με μεγάλη υπέρβαση των οριακών τιμών που καθορίζονται στην νομοθεσία. Τα βασικά προβλήματα που αναφέρονται και στις ε, αναφορές και που αφετέρου ε, διαπιστώσαμε και εμείς μέσω της ανάλυσής μας είναι φυσικά η κυκλοφορία, η κυκλοφορική συμφόρηση στις πόλεις, αλλά και το είδος των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στις πόλεις. Το βασικό πρόβλημα σε σχέση με την ποιότητα του αέρα ε, προφανώς πηγάζει από τα οχήματα diesel γιοταχή αλλά και επαγγελματική χρήση αυτοκίνητα. Η ατμοσφαιρική ρήπη είναι κατά βάση τα PM10, το διοξείδιο του αζότου. Σε κάποιες περιοχές και πόλεις υπάρχει πρόβλημα με το όζον και σε κάποιες περιοχές και πόλεις υπάρχει και πρόβλημα με το βενζοπυρένιο. Στην Ισπανία επίσης έχει υπάρξει μια συζήτηση σχετικά με την τοποθεσία στην οποία βρίσκονται οι σταθμοί παρακολούθησης που σε αρκετές περιπτώσεις έχουν μεταφερθεί λόγω της εφαρμογής ε, της οδηγίας 2008 κάθετος 50. Αντίστοιχη συζήτηση έχει υπάρξει και στις, έχει υπάρξει στις Βρυξέλλες λόγω της, μετακο, με, της μεταφοράς κάποιου σταθμού παρακολούθησης ε, σε άλλο σημείο εντός της πόλης λόγω κατασκευαστικών έργων. Το εξετάζει ακόμη και το ελεκτικό συνέδριο αυτό το, αυτή την υπόθεση. Επίσης, γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό νέων, ε, της κατασκευής νέων οδικών αξώνων. Είναι προφανές ότι οι νέοι δρόμοι θα δημιουργήσουν ακόμη περισσότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση, τα έργα ακόμα περισσότερο βεβαίως, και αυτό θα επιδεινώσει έτσι περαιτέρω την ποιότητα του αέρα στις πόλεις. Λοιπόν, τα προβλήματα πάντως είναι παρόμοια σε όλη την Ευρώπη. Δεν υπάρχει κάτι που να διακρίνει τη μία πόλη από την άλλη. Παρόμοια προβλήματα, ξαναλέω, είναι τα, τα ε, σε όλες τις πόλεις. Εκτός από τη Λομβαρδία, που αποτελεί εξαίρεση, είναι μεγάλη περιφέρεια, με μεγάλο πληθυσμό και εκεί υπάρχει πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τους ατμοσφαιρικούς ρήπους. Αυτό που κάναμε στη συνέχεια ήταν να εξετάσουμε τις βέλτιστες πρακτικές και αυτό που είδαμε ότι υπήρχαν αρκετά παραδείγματα αλλά και πρωτοβουλίες, projects των πολιτών που δείχνουν ξεκάθαρα ότι πολλές πόλεις έχουν προσπαθήσει να βρουν λύσεις για να καλυτερεύσουν την ποιότητα της ζωής των κατοίκων και αυτό που είδαμε και υπογραμμίζουμε στη μελέτη μας είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ενσωματωμένη πολιτική σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις που λαμβάνει υπόψη της τα δημόσια μέσα μεταφοράς, μαζικής μεταφοράς μέσα βιώσιμης ανάπτυξης, πώς μπορεί κανείς να περπατάει περισσότερο, να χρησιμοποιεί το ποδήλατο, καλύτερη χρήση τεχνολογίες που αφορούν τα οχήματα αλλά και τα καύσιμα, πολιτικές που αφορούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους όλα αυτά. Πιο συγκεκριμένα και σε σχέση με την ποιότητα του αέρα, βέλτιστες πρακτικές είναι οι ακόλουθες, ζώνες χαμηλών εκπομπών, αναδιανομή του δημόσιου χώρου, τόσο ώστε να μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί ποδήλατα και να, περπατεί, να περπατάει πιο εύκολα, διάφορα σχήματα σε ό,τι αφορά την φορολόγηση του ντίζελ κτλ. Επίσης, ό,τι αφορά τα λιμάνια, αλλά και τα φορτηγά. Ναι, Πολιτικές, ούτως ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε την μόλυνση από αυτά. Η χρήση της θέρμανσης πολύ συχνά έχουμε να κάνουμε με χρήση άνθρακα Ένα ζήτημα που επίσης ενισχύει τη μόλυνση. Για παράδειγμα τα κτίρια που δεν έχουν αναπαλαιωθεί. Παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών είναι στη διάθεση του κοινού. Για παράδειγμα καλύτερη συντήρηση αναπαλαίωση των κτίριων, πολύ σημαντικό, για να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των συστημάτων αυτών θέρμανσης, αλλά και η απαγόρευση συγκεκριμένων καυσίμων, όπως είναι ο άνθρακας, για παράδειγμα. Αυτό ισχύει στο Δουβλίνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε ό,τι αφορά τώρα την γεωργία. Η ένα στοιχείο της γεωργίας που δεν συμβάλλει και τόσο πολύ στην μόλυνση του αέρα είναι οι εκπομπές αμμονίας. Επίσης, η καύση, η καύση ζυζανιοκτώνων μπορεί επίσης να συμβάλλει στη μόλυνση του αέρα, άρα θα πρέπει να απαγορευτεί ως πρακτική. Επίσης θα πρέπει να α, μειωθεί η χρήση αμμονίας. Σε ό,τι αφορά τις κατασκευές τώρα, αυτό είναι ένα ζήτημα για τις μεγάλες πόλεις, ιδίως σε ό,τι αφορά της που όπου υπάρχει ιδιαίτερη κατασκευαστική δραστηριότητα. Συμβαίνει και στην Αυστρία, στη, στη δική μου τη χώρα. Υπάρχουν περιοχές όπου οι εκπομπές ρήπων από την κατασκευαστική δραστηριότητα έχει μειωθεί υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες, ε, καθώς επίσης και για τη μείωση ε, της κυκλοφορίας σε περιοχές όπου υπάρχει κατασκευαστική δραστηριότητα. Πολλά μπορούν να γίνουν και σε αυτό το τομέα. Όπως επίσης, όπως για παράδειγμα τα φίλτρα για το πετρέλαιο. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι πολλά από τα μέτρα δεν χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα, αλλά για παράδειγμα να, να βελτιώσουν την, την ενεργειακή αποδοτικότητα, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ποιότητα της ζωής, την δημόσια υγεία, να ενδυναμώσουν το σκεπτικό των λεγόμενων smart cities. Όλα αυτά, όλες αυτές οι βέλτιστες πρακτικές, όλες αυτές οι διαφορετικές στρατηγικές αλληλοσυμπληρώνονται. Και όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας όταν προσπαθούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με το τι θα είναι πιο αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση των ε, προβλημάτων. Τέλος, πρέπει να υπάρχει ισχυρή δημόσια και πολιτική στήριξη για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Υπάρχουν παραδείγματα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχεδόν τελειώνει η παρουσίασή μου. Αυτό που προτείνουμε για τις πόλεις που είδαμε είναι αυτά τα παραδείγματα των, των ζώνων χαμηλής εκπομπής, των ζώνων χαμηλής εκπομπής, να μπορέσουμε να προωθήσουμε τους ποδηλατόδρομους, τους α, πεζόδρομους, καλύτερη διαχείριση όλων αυτών των εναλλακτικών μέσων μετακίνησης σε ό,τι αφορά τώρα την καύση ξύλου, είναι πολύ σημαντικό να μειωθεί σε περιφερειακό επίπεδο, κάτι το οποίο θα βοηθήσει με τη σειρά του την ποιότητα του αέρα στις πόλεις Είναι επίσης πολύ σημαντικό να παρακολουθούμε την εφαρμογή, να παρακολουθούμε την πρόοδο όλων αυτών των μέτρων, να υπάρχει ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα, να είναι ξεκάθαρες και οι ευθύνες. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρος. Έχει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you very much. Uh, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την Επιτροπή σας που προβάλλει αυτό το ζήτημα γιατί είναι πάρα πολλές οι αναφορές ακριβώς όπως ξέρετε. Ε, αυτό σημαίνει το πόσο ενδιαφέρονται οι Ευρωπαίοι για το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης και μόλυνσης. Και να υπενθυμίσουμε ότι πέραν των 7 πόλεων που κάλυψε αυτή η μελέτη έχουμε γύρω στις 130 πόλεις στην Ευρώπη που δεν έχουν ε, το στάνταρ το οποίο έχουμε ορίσει στην Ευρώπη και αυτό αφορά και τα, διοξίδια, τα οξύδια του αζότου και άλλες ουσίες Έχετε πάρα πολλές πηγές ε, ε, για αυτή τη μελέτη. Είχαμε όλα τα δεδομένα από παντού. Έχουμε επίσης ε, τον έλεγχο των σχετικών πολιτικών από το ελεγκτικό συνέδριο. Τα καλύψε τελευταία. εμείς. Έχουμε τώρα να πούμε μερικά πράγματα. Έχουμε να σταθούμε σε κάποια ζητήματα για τις τάσεις που αναφέρατε και εκεί επιφυλασσόμαστε. Λέει η μελέτη, όχι η προφορική παρουσίαση, ότι για τις Βρυξέλλες δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε μια ε, σαφή καθοδική τάση για τις εκπομπές του αζότου και για το Μιλάνο, όχι αναγκαστικά για την περιφέρεια της Λομβαρδίας, ότι εκεί πέρα επίση υπάρχει βελτίωση της κατάστασης, αλλά εμείς έχουμε πούμε ότι οι εκπομπές ε, ε, του αζότου είναι σχεδόν 50% πάνω από τις οριακές τιμές και όπως είπατε και εσείς ε, έχουμε δύο ή τρεις φορές πάνω από το όριο ε, εκπομπές ε, αυτό είναι συναγερμός. Θα πρέπει να γίνουν πολλά σε αυτό το τομέα να εξασφαλίσουμε ότι ο κόσμος μπορεί, μπορεί να ανασάνει καθαρό αέρα. Ε, επίσης να υπενθυμίσουμε ότι η νομοθεσία εφαρμόζει την αρχή της επικουρικότητας σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή να επιλέξουν τα κράτη-μέλη τα μέσα πολιτικής για το πώς καλύτερα θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σε κάθε επίπεδο. Πάντως, οι μελέτες έτσι και είναι χρήσιμες γιατί δείχνουν ότι υπάρχουν τα μέσα. Μπράβο επομένω που είπατε ότι χρειάζεται ολοκληρωμένη προσέγγιση. Και δεν είναι μόνο τα μέτρα για την καθαρή ατμόσφαιρα, αλλά υπάρχουν και μέτρα για ενεργειακή αποτελεσματικότητα, μεταφορές, γεωργία, κλίμα, Όλα αυτά ωφελούν την καθαρή ατμόσφαιρα. Ευχαριστούμε που μας είπατε τη γνώμη σας, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι αυτός ο διάλογος θα μας ε, δώσει πολλές ιδέες. Θέλει κανείς το λόγο. Πάντως ευχαριστούμε εσάς κύριε για τη μελέτη για την παρουσίασή σας. Α, κάποιος δει το λόγο. Η κυρία Βαλίνα, έχετε το λόγο, δεν σας είδα, συγγνώμη. Ήθελα να σας ρωτήσω, μια που μας μιλήσατε για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και άλλα πολλά, που κατέληξε η στο πώς επηρεάζουν την κατάσταση τα αεροπλάνα, τα ε, αεροδρόμια, γιατί εγώ ξέρετε προέρχομαι από κάποιο μεγάλο λιμάνι και νομίζω ότι υπάρχουν εκπομπές από τα σκάφη, από τα πλοία και πολλές φορές αποθηκεύονται διάφορες ουσίες, ε, έταλα διάφορα στα λιμάνια και αυτά επίσης μολύνουν. Έχουμε επίσης ε, τους λέβητες, τους καυστήρες για τα αποτεφρωτήρες τέλος πάντων για τα σκουπίδια. Όλα αυτά τα λάβατε υπόψη για τη μελέτη σας. Έχετε το λόγο, λέει ο Πρόεδρος, στον εισηγητή. Ναι, ναι. Λάβουμε υπόψη τις διαφορετικές αιτίες της μόλις της ατμόσφαιρας. Κυρίως για τις πόλεις. Ναι, λάβουμε υπόψη τον ρόλο των πλοίων. Έχουμε μια αξιόλογη τέτοια μελέτη. Και υπάρχουν και σχετικές προτάσεις για το τι να κάνει κανείς για τις εκπομπές των πλοίων στα λιμάνια. Τώρα αφορά τα αεροπλάνα, δεν το κοιτάξαμε συγκεκριμένα το θέμα, αλλά βέβαια Έχουμε μέτρα για τις ε, δημόσιες μεταφορές και γενικά τρέτα. Την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, οπότε λαμβάνουμε υπόψη και αυτές τις... Α, ξέχασα να σας ρωτήσω κύριε Βαλίνα. η βιομηχανία δεν έχει συνέπειες. Σε κάποιες ε, πόλεις υπάρχουν εργοστάσια μέσα στην πόλη, τέλο πάντων στα προάστια και ούτε εκεί λαμβάνονται από όλους τα μέτρα που θα έπρεπε. ο εισηγητής. Δεν αναφέραμε τα εργοστάσια, αλλά έχετε δίκιο. Σε κάποιες πόλεις υπάρχει μια τέτοια κατάσταση με εργοστάσια. Δεν μπορούμε να γενικεύσουμε όμω τα συμπεράσματα. Δώσαμε γενική άποψη των πραγμάτων. Ε, θα πρέπει κανείς περιπτωσιολογικά να το εντοπίσει το πρόβλημα. Και υπάρχει και η οδηγία για τις εκπομπές της βιομηχανίας που πρέπει να εφαρμοστεί παντού στην Ευρώπη, για όλα τα εργοστάσια. Και θα πρέπει να, να συμμορφώνονται οι βιομηχανίες με αυτήν την οδηγία. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση και για τη μελέτη. Είναι κορυφαία πολιτική προτεραιότητα. Είμαστε μία από τι τρει χώρε στι οποίε αναφερθήκατε όσον αφορά τα οξύδια του αζότου. Στη Βρετανία. Όλο ένα και περισσότεροι ανησυχούν. Είπαμε ότι έχουμε πάνω από 2.000 ε, σχολεία που βρίσκονται σε πάρα πολύ μικρή απόσταση από ε, βιομηχανίε. Το θέμα είναι καυτό πολιτικά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι άριστες πρακτικές σε εθνικό επίπεδο. Να δούμε δηλαδή τι διαφορά στην αντιμετώπιση υπάρχει από χώρα σε χώρα. Γιατί στη χώρα μας συζητείται ακριβώς το θέμα της αδράνειας από πλευρά του κράτους. προσεχούμε ιδίω τι γίνεται σε περιφερειακό δημοτικό επίπεδο. Όλη η νομοθεσία είναι νομοθεσία ευρωπαϊκή και στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα. Ψηφίσαμε για τις εκπομπές των αυτοκινητών νέους κανόνες. Οπότε και σας ερωτώ, εντοπίσατε τίποτα κενά, παραθυράκια που θα πρέπει να διορθωθούν στο επίπεδο κοινωτικού δικαίου να καθισκάσουν την ανησυχία του κόσμου για την ρήπανση. Τέλος πάντων θα πρέπει να εφαρμοστεί και το ισχύον δίκαιο πλήρω. Και βέβαια θα πρέπει να συνοηθούμε με όλες τις αναμόδιες επιτροπές περιβάλλοντος, μεταφορών, εδώ στο Κοινοβουλίο. Ο Πρόεδρος. Κυρία Εύη. Και μετά εσείς κύριε Σίγητα. Κυρία Εύη. Σας ευχαριστώ και εγώ, Πρόεδρε, και τον εισηγητή για την ενδιαφέρουσα μελέτη σήμερα. Είναι πολύ σημαντική μέρα γιατί σήμερα στο Συμβούλιο, στο Συμβούλιο πρόκειται να γίνει ψηφοφορία όσον αφορά την θέση του Συμβουλίου για τον νέο κανονισμό, για τον περιορισμό τον εγωμό διοξιδίου από φορτηγά και αυτοκίνητα. θα πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες που σήμερα που προσπαθούν να κάνουν κάτι για το κλίμα, για την υγεία. Τα πράγματα βέβαια ακόμα είναι αβέβαια για το θέμα. Πέστε μας, οι επιστήμονες στις μελέτες δεν λένε ότι θα πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές. Έτσι να προστατεύσουμε το κλίμα, έτσι να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις του Παρισιού. Διάβησα. Εκεί που λέτε πρέπει να γίνει 50, 60, 70% ε, μείωση μέχρι το 2030. Όλα αυτά τα προσκεφθήκαμε στο Παρίσι. Το κοινοβούλιο λέει 40% μείωση. Και για πέστε μας, άρκουν αυτά Αυτά θα προστατεύσουν την υγεία των Ευρωπαίων. Έτσι θα έχουμε μια κινητικότητα καθαρή στην Ευρώπη. Και άλλα βέβαια αυτός από την υγεία θα πρέπει να μην ξεχνάμε και την απασχόληση στην Ευρώπη. Okay, thanks a lot. Maybe first, uh, Ωραία. Για το πρώτο ερώτημα σχετικά με την εθνική νομοθεσία και τη δική μας ε, νομοθεσία, την ευρωπαϊκή δηλαδή. Στην πολύ μικρή έκταση ε, μελέτη που εκπονήσαμε, προφανώς δεν μπορέσαμε να εξετάσουμε όλο το εύρος των νομοθεσιών που αφορούν τα οχήματα, ε, ούτε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένε προτάσεις. Θα ήταν κάτι υπερβολικό αυτός αξίωση βεβαίως και από τον εαυτό μας. Βεβαίως, σίγουρο είναι ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, φορολογία των οχημάτων diesel, των καυσίμων diesel. Αυτά βεβαίω αναπόκεινται στι εθνικές κυβερνήσεις να τα αποφασίσουν. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι φυσικά πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι τα μελλοντικά οχήματα πράγματι θα συμμορφώνονται με τις ε, οριακές τιμές εκπομπών. Αυτό είναι σίγουρα πολύ σημαντικό. Και βεβαίως χρειάζεται να παρασχεθεί και ένα πλαίσιο το οποίο θα διευκολύνει και θα επιτρέπει την μετάβαση σε ένα νέο σύστημα μεταφορών φιλικό προς το περιβάλλον. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να υποστηριχθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά το ερώτημα που σχετιζόταν με τις δεσμεύσεις των Παρισίων και τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή. Βεβαίως, όλα αυτά τα στοιχεία βοηθούν με την ε, μοναδική εξαίρεση της καύσης βιομάζας για οικιακή χρήση. Αλλά στην, ε, στην περίπτωση των οχημάτων ε, υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση προς τον εξηλεκτρισμό, προς την διάδοση και την προώθηση συστημάτων δημόσιας συγκοινωνίας, ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου ε, και αυτά όλα βοηθούν και στην επίτευξη των στόχων του Παρισιού και στην, στο στόχο της βελτίωσης του, της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Σας συγχαίρουμε για το εξαιρετικό σας έργο και την μελέτη που μας παρουσιάσατε. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, περνάμε τώρα ε, στα υπόλοιπα θέματα. Έχουμε τρία από την ε, Βουλγαρία αναφορές που αφορούν την πόλη Στάρα Ζαγόρα. Υπάρχουν και εκεί προβλήματα με τη ρήπανση του αέρα. Οι αναφέροντες είναι παρόντες, όχι. Από ό,τι βλέπω. Τότε θα ήθελα να ζητήσω το, από τον κύριο Μίκε να τοποθετηθεί όσον αφορά τη συγκεκριμένη αναφορά. Ευχαριστώ πολύ. Η αναφορά αυτή αφορά την ε, ποιότητα του αέρα και τα σχετικά προβλήματα στη Σταραζαγόρα. Κάτι το οποίο προκλήθηκε και από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης. Με βάση την συνθήκη προσχώρησης του 2007 πολλές εγκαταστάσεις καύσης είχαν λάβει εξαίρεση όσον αφορά την εφαρμογή των οριακών τιμών που προβλέπονται στην Εθνική Νομοθεσία για τη Βιομηχανία. Οι εξαιρέσεις αυτές ίσχυσαν έως το τέλος του 2014, το αργότερο. Και ε, είχαν προβλεφθεί ώστε να δοθεί αρκετός χρόνος για να γίνει η αναβάθμιση αυτών των εγκαταστάσεων προκειμένου να μπορούν να τηρούν τις, ε, τα όρια της, Ευρωπαϊκή ε, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ε, είχαν οριστεί ευρωπαϊκά και εθνικά ανώτατα όρια και εκεί φαίνεται να υπάρχει η πρώτη παραβίαση. Η Κομισιόν λοιπόν ξεκίνησε τη διαδικασία επί το 2011 και έπειτα από πολλές Επαφέ, με τις βουλγαρικές αρχές αποφάσισε εξετάζοντα την περίπτωση το 2015 να κλείσει τη συγκεκριμένη υπόθεση διότι τα εθνικά όρια αφενό βάσει της ε, συνθήκης προσχώρηση, δεν ίσχυαν πλέον και επειδή η Κομισιόν ερεύνησε την υπόθεση των ε, επιμέρους εγκαταστάσεων καύσης και δεν διαπίστωσε πουθενά παραβίαση των ε, ορίων βιομηχανικής προέλευσης. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εξέτασε το ζήτημα της ποιότητας του αέρα με βάση την οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και εκεί έχει ξεκινήσει η διαδικασία παραβάσει εναντίον της πόλης της Στάρας Αγόρα για την ε, ε, υπέρβαση των ορίων PM10 και διοξιδίου του θείου. Η διαδικασία αυτή οδήγησε σε απόφαση του δικαστηρίου τον Απρίλιο του 2017 και η Κομισιόν παρακολουθεί στενά την ε, εφαρμογή από πλευρά Βουλγαρία τη απόφαση αυτή του δικαστηρίου όσον αφορά τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προκειμένου να τηρούνται τα ε, όρια και οι εκπομπέ ε, στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Αν αποδειχθεί ότι τα μέτρα δεν, ε, που έχουν ληφθεί από τις βουλγαρικές αρχές δεν επαρκούν, ενδέχεται να αναλυθούν περαιτέρω νομικές δράσεις. Ευχαριστώ πολύ. It is really a very good coincidence, this petition... Είναι σύμπτωση ότι η αναφορά αυτή σχετίζεται και με την παρουσίαση που μόλις παρακολουθήσαμε. Εγώ θέλω να σας πω ότι πριν από δύο εβδομάδες ήμουν στη Στάρα Ζαγόρα. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό, είναι πραγματικό. Οι πολίτες περιμένουν οποιαδήποτε βοήθεια, πρέπει να σας πω, γιατί το πρόβλημα ε, χρονίζει. Μάλιστα, πολλές φορές αναφέρεται και στον ε, τύπο της ε, Βουλγαρίας. Είναι ένα πολύ αναγνωρίσιμο πρόβλημα, λοιπόν, στην Βουλγαρία υπάρχουν ακόμη και δημόσιες διαμάχες για το ποιος ευθύνεται για την κατάσταση, γιατί υπάρχουν κάποιες υποψίες από διάφορες πηγές. Να συνοψίσουμε όμως και οι τρεις αναφορές αφοράν την σημαντική ρήπανση του ατμοσφαιρικού αέρα γύρω από τη Στάρα Ζαγόρα και το βασικό πόρισμα είναι ότι υπάρχουν βαρέα μέταλλα και χημικές ουσίες σε φυτά, αέρα και τρόφιμα. Αυτό θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία του πληθυσμού. Οι αναφέροντε λοιπόν και στι τρει αυτέ τι αναφορέ, διότι είναι τρει διαφορετικοί ε, αναφέροντε και οργανώσει από πίσω, ισχυρίζονται ότι οι αρμόδιες βουλγαρικές αρχέ δεν έχουν καταφέρει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στι 5 Απριλίου απεφάνθη ότι η Βουλγαρία δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την, ε, τον σεβασμό των οριακών τιμών για το PM10 και δεν κατάφερε να ε, υποβάλει ένα σχέδιο μέτρων τα οποία θα ε, κρατούν τις εκπομπές στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Οι υπηρεσίε της Κομισιόν λοιπόν τώρα βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τις βουλγαρικές αρχές ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Κάποια πράγματα λοιπόν έχουν κλείσει αλλά κάποια πράγματα παραμένουν ανοιχτή, ανοιχτά. Η συνεργασία συνεχίζεται και μπορώ να σας πω και από προσωπική εμπειρία ότι όποτε δημοσιεύεται ένα τέτοιο ε, και παίρνει διαστάσεις στην κοινή γνώμη ε, ένα τέτοιο περιβαλλοντικό πρόβλημα, ε, οι τοπικές αρχές ξαφνικά γίνονται πιο συνεργάσιμες. Και δεδομένου ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει τις συνεργασίες της και τις επαφές της με τις βουλγαρικές αρχές, εγώ θα συνιστούσα να τις κρατήσουμε ανοιχτές τις αναφορές αυτές και αναλαμβάνω προσωπικά την ευθύνη να σα ενημερώνω για την πρόοδο. Γιατί κάποιε φορέ, ξέρετε, δεν χρειάζεται να γίνονται διερευνητικέ επισκέψει. Μπορεί να πάει και ένα ευρωβουλευτή προσωπικά και να ελέγξει τι συμβαίνει επί τόπου. Θα είναι λοιπόν εξαιρετικό το μήνυμα που θα αποστείλουμε αν αφήσουμε τις αναφορές αυτές ανοιχτές ώστε να βοηθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας αυτή τη συνεργασία, αν θέλετε, μεταξύ Κομισιών και Βουλγαρικών Αρχών. Ευχαριστούμε πολύ. Χαίρομαι που η Επιτροπή κατανοεί το πρόβλημα και έχει αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες Ε, βεβαιω εκκρεμεί ακόμη το θέμα, είναι ανοιχτό. Όπως συζήτησε ο συνάδελφο, θα, ζητήσουμε, θα κρατήσουμε ανοιχτή αναφορά και θα στείλουμε μια επιστολή στη βουλγαρική κυβέρνηση και έτσι θα πούμε ότι εμείς ε, παρακολουθούμε προσεκτικά την εξέλιξη. Αν συμφωνείτε, τότε θα αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά ή τις αναφορές. Η επόμενη αναφορά προέρχεται από την Πολωνία. Αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ατμόσφαιρας για τη χώρα. Δεν παρίσταται ο αναφέρον. Θα δώσουμε το λόγο. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στην Πολωνία. Ζητεί ο αναφέρον να πιεστεί η κυβέρνηση να βελτιώσει την ποιότητα της ατμόσφαιρας όσον αφορά την κυκλοφορία των οχημάτων, και την θέρμανση των κατοικιών ως αιτίε της επιδείνωσης. Ε, το Ευρωπαϊκό Διαστήριο έχει ήδη καταδικάσει τη χώρα φέτος γιατί δεν σεβάστηκε η χώρα, δεν ετήρησε τις οριακές τιμές που προβλέπονται από τη σχετική οδηγία γιατί δεν λήφθησαν τα δέοντα μέτρα ε, στον προγραμματισμό της. Και επίσης γιατί δεν μετέφερε σωστά τη σχετική οδηγία στο ιστορικό δίκαιο. Επίσης, το οξύδιο του αζότου και για αυτή την ουσία το 2016 η Ευρωπαϊκή Επίτροπη απίθυνε όχληση προς την κυβέρνηση ότι δηλαδή αυτή η ουσία έχει υπερβεί τις οριακές τιμές που προβλέπονται και ε, για το ότι η χώρα δεν επεξεργάστηκε κάποιο σχέδιο αντιμετώπιση του προβλήματος. Το Σεπτέμβριο φέτος, πριν από μία εβδομάδα δηλαδή, η Επιτροπή ειδοποιήθηκε από την Πολωνία για το τι στοιχεία υπήρχαν το 2017. Οπότε τώρα με τα στοιχεία που έχουμε θα αξιολογήσουμε συνολικά το τι γίνεται στη χώρα. Να δούμε επομένω αν συντρέχει περίπτωση παραβίαση του δικαίου. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ θετική η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νομίζω ότι θα βοηθήσουμε αν κρατήσουμε αυτή την αναφορά. Θα περιμένουμε επομένω τα αποτελέσματα της αναλυσής σας. Και στη συνέχεια θα δούμε αν συμφωνούμε για το τι θα γίνει. Τώρα έχουμε άλλες δύο αναφορές από το Φράιμπουργκ και από το Αμβούργο. Έχουν ε, σύναφες, θέμα αυτές οι δύο αναφορές που θα εξεταστούν στη συνέχεια και σε αυτές τις αναφορές θίγεται το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος και οι σχετικές ε, παραβάσεις του νόμου. Αν δεν κάνω λάθος, δεν παρίστανται οι αναφέροντες. Ας το λόγο στον Νικόλα Όστερτα, που είναι ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως αναφέρατε, η αναφορά 1083 σε ό,τι αφορά τα ανώτατα όρια του μονοξιδίου του άνθρακα στην περιοχή Φράιμπορκ, στην επαρχία Μπράισκαου της Γερμανίας και η αναφορά 1363 του 2015 επίσης για την ποιότητα του αέρα στο Αμβούργο και οι δύο αναφορές υπογραμμίζουν την αδυναμία των ε, ηθήνοντων να αναλάβουν δράση. Οι παρατηρήσεις μας, όπως ε, αναφέραμε και σήμερα το πρωί, η Επιτροπή αποφάσισε να καταγγείλει την ε, Γερμανία καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μην συμμόρφωση με τα ανώτατα ωραία εκπομπής μονοξυδιού του άνθρακα. σε ό,τι αφορά τις ζώνες του Φράιμπουργκ και του Αμβούργου, σε το αφορά την περίπτωση της Γερμανίας. Σύμφωνα με την αναφορά που παρήχε η Γερμανία, την τις αναφορά για την ποιότητα του αέρα τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε, η συγκέντρωση μονοξιδίου του άνθρακα ήταν 49 ενώ το 2000 ήταν 9 ε, μικρογραμμάρια, δηλαδή περισσότερο από το ανώτατο επιτρεπτό όριο. Για το Αμβούργο η τιμή ήταν 58 μικρογραμμάρια, δηλαδή 18 γραμμάρια, μικρογραμμάρια, με συγχωρείτε, πάνω από το επιτρεπτό όριο. Έχουμε δηλαδή μία α, παρέκβαση της τάξης του 45% από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια. Τέλος θα ήθελα να σημειώσω την πρόσφατη ανακοίνωση από τον αναφέροντα σύμφωνα με τον οποίο μας ενημερώνει για τα μέτρα που λαμβάνουν οι κάτοικοι στην περιοχή του Φράιμπορκ ή Κομισιόν παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις πρωτοβουλίες των πολιτών, των κατοίκων σε σχέση με την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα. Παρόλα αυτά σημειώνουμε ότι οι πρωτοβουλίες αυτές δεν ε, μπορούν να επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα σε σχέση με τα επιτρεπτά όρια. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και όταν δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι, τα μέτρα που λαμβάνουν οι ίδιοι οι κάτοικοι και η δραστηριότητά τους μας δίνουν σημαντικά στοιχεία για το πώς λειτουργούν οι ίδιοι οι κάτοικοι και μπορούν επίσης να αυξήσουν και την επίγνωσή μας σε σχέση με την κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό που θέλω να συγκρατήσω είναι ότι η θέση της Επιτροπής σε Γενικές Γραμμές είναι θετική. Ενεργά εξετάζουν την αναφορά αυτή και εργάζονται από κοινού με τους αναφέροντες κάτι το οποίο ισχύει και για την προηγούμενη αναφορά αυτό που έχω να προτείνω λοιπόν είναι να περιμένουμε μέχρι η Επιτροπή να τελειώσει τη δουλειά της να κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή και να δράσουμε στη συνέχεια ανάλογα. Ευχαριστώ. Äh, Δεν θα ήταν σωστό να μην ασχοληθούμε και με την επόμενη αναφορά που έρχεται από τη Γαλλία, Γάλλος υπήκος είναι ο αναφέρον, έχει να κάνει με την καλύτερη ποιότητα του αέρα. Ο αναφέρον δεν είναι παρόν και πάλι θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, τον κύριο Μιγέλ Ντε Χουαρές. Έχετε το λόγο κύριε. Πολύ καλά, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρόκειται για μία αναφορά που είναι ήδη αρκετά παλιά. Έχει να κάνει με την οδηγία της καλυτέρευσης του αέρα σε σχέση με τις εκπομπές και επικρίνει την δράση της Γαλλίας σε προσημόρφωση της οδηγίας αυτής. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η Κομισιόν μέχρι στιγμής δεν έχει θεωρήσει θεμητό να επανεξετάσει την συγκεκριμένη οδηγία. Έχουν γίνει κάποιες μικρές τροποποιήσεις ό,τι αφορά τους πίνακες. Η Κομισιόν εφαρμόζει την οδηγία αυτή. Σε κάθε περίπτωση όμως η Κομισιόν έχει επανεξετάσει την εφαρμογή της οδηγίας, το λεγόμενο fitness check, με στόχο να δει πώς έχει λειτουργήσει την τελευταία δεκαετία η εφαρμογή της οδηγίας. Έχει συγκρίνει τους στόχους που είχαν τεθεί, αλλά και αυτούς που επιτεύχθηκαν. ούτω ώστε να μπορέσει να βελτιωθεί η αποδοτικότητα, αλλά και να επιτευχθούν βεβαίως οι στόχοι, που βεβαίως είναι η καλυτέρευση της ποιότητας του αέρα και οι επιπτώσεις της στην υγεία των ανθρώπων, αλλά και στο περιβάλλον. Η αξιολογήσεις αυτές έγιναν με την συμμετοχή των κρατών μελών, με κάθε διαφάνεια αλλά και με, με τη συμμετοχή διαφόρων οργανώσεων και υπήρξε και μια δημόσια διαβούλευση. Σε κάθε περίπτωση η Κομισιόν επισυνάπτει ιδιαίτερη σημασία α, των διαφορών που επισημαίνουμε στα κράτη-μέλη. Χρησιμοποιούμε μια σειρά από μέτρα και δίκτυα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε ποιες είναι οι ιδιαίτερες δυσκολίες σε κάθε κράτος μέλος και να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα, ούτως ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συμμόρφωση. Αυτό ισχύει σε γενικέ γραμμέ ό,τι αφορά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τον ειδικό διάλογο σε ό,τι αφορά την καλυτέρευση του αέρα, το λεγόμενο Clean Air Dialogue. Η Κομισιόν ενθαρρύνει επίσης και τα διάφορα εθνικά μέσα, ούτως ώστε να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να εξετάζουν κατά πόσο η εφαρμογή της οδηγίας γίνεται ορθά. Η Κομισιόν επίσης έχει ξεκινήσει διαδικασίες εναντίον 16 κρατών μελών γιατί ξεπερνούν τα ανώτατα επιτρεπτά μέτρα τα οποία με την εξαίρεση ενός και μοναδικού κράτους βρίσκονται στα πρόθυρα μιας, κατασ... μιας καταγγελίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αναφέρομαι στην Βουλγαρία και την Πολωνία. Με την εξαίρεση, με συγχωρείτε, της Πολωνίας και της Βουλγαρίας, οι οποίες πρόσφατα έδειξαν στοιχεία βελτίωσης. Η Ουγγαρία, η Ιταλία και η Ρουμανία τον τελευταίο χρόνο οδηγήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σε ό,τι αφορά το μονοξίδιο του άνθρακα, τώρα 13 κράτη-μέλη έχουν παραβιάσει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια, μεταξύ των οποίων τρία, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, έχουν ξεπεράσει τα όρια και έχουν οδηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης. Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι την Γαλλία τώρα. Ο αριθμός των ε, βλαβερών σωματιδίων ε, πέρασε από το 2015 στο 2017 από 10 σε 3, αλλά παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Πιο συγκεκριμένα, τα βασικότερα αστικά κέντρα της χώρας εμπλέκονται. Πρώτα απ' όλα, το Παρίσι, όπου η παρουσία τέτοιων σωματιδίων είναι διπλάσια από το ανώτοτο επιτρεπτό όριο. Στη Μασαλία τα πράγματα δεν είναι πολύ καλύτερα. Επίσης, ένας ε, τέτοιου τύπου νούμερα ε, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου σαν μέτρα που θα πρέπει να λάβουμε άμεσα. παρά την προειδοποίηση που εστάλθη η γαλλική κυβέρνηση στις 10 Ιουλίου του 2017 και την ανάγκη δημιουργίας ενός σχεδίου για την καλυτέρευση του αέρα και την τήρηση του επίπεδου του διξιδίου του άνθρακα σε αποδεκτά επίπεδα. Τα μέτρα δεν ήταν αρκετά γιατί εξακολουθούν να υπερβαίνουν τα όρια. Ως εκ τούτου, η Κομισιόν αποφάσισε να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έναντι συμπεράσματος, η Κομισιόν, σε σχέση πάντοτε με την οδηγία για την καλυτέρευση του αέρα, βάση συγκεκριμένων ενεργειών, ενεργεί εναντίον της Γαλλίας η Κομισιόν αποφάσισε να αναλάβει δράση εναντίον της Γαλλίας για μη συμμόρφωση με τη συγκεκριμένη οδηγία. Ο Πρόεδρος. Να σας ευχαριστήσω που μας είπατε τις απόψεις σας και ευχαριστούμε επίσης που ασχοληθήκατε με το πρόβλημα. Ε, αξίζει πάντως ε, κανείς να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για αυτή την υπόθεση. Σύμφωνα με όσο μας είπαν οι ειδικοί, θα πρέπει να κρατήσουν αυτή, την αγορά και να περιμένουν να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Κύριε Γιάρα. Ναι, συμφωνώ. Απλά θέλω να κάνω μια γενική παρατήρηση για όλες τις αναφορές. Λοιπόν, θεωρώ δεδομένο ότι οι αρκετές τιμές που είχαν αποφασιστεί για τη βελτίωση του ατμοσφαιρικού αέρα ε, αποφασίστηκαν και με τη συμμετοχή των κρατών μελών. Εδώ μάλλον ισχύει και αυτή η ρίση που χρησιμοποιώ πολύ συχνά. Το θέμα δεν είναι να βελτιώσουμε τις, ε, τα στατιστικά στοιχεία, αλλά την πραγματικότητα. Και φαντάζομαι ε, ότι έχουμε να κάνουμε για άλλη μια φορά με μια περίπτωση όπου τα κράτη-μέλη συνεφώνησαν ως προς τις οριακές τιμές στα χαρτιά, δεν κάνουν τίποτα όμως ή τέλος πάντων κάνουν ελάχιστα όσον αφορά την εφαρμογή. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, πολύ συχνά στη συνέχεια ε, ακούγονται απόψεις από τα κράτη-μέλη ότι μας επιβάλλονται αυτά τα όρια από τις Βρυξέλλες κτλ. Λοιπόν, όχι. Είναι ευθύνη των κρατών μελών, έστω και καθυστερημένα, να αναλάβουν μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης. Γι' αυτό και ε, αφήνουμε ανοιχτά Ανοιχτέ τι αναφορές αυτές. Δεν είναι καπρίτσιο των Βρυξελών. Όποιο αποφασίζει εδώ στα όργανα συνομοθέτηση συγκεκριμένε οριακές τιμέ, έχει συνέχεια ευθύνη να τα εφαρμόσει και όλα αυτά τα μέτρα. Ε, Δυστυχώ, πολλέ φορές η διαδικασία αυτή είναι επίπονη, δεν πειράζει όμως. Αυτό πρέπει να μας δίνει θάρρος και στις ε, ε, μελλοντικές νομοθετικές διαδικασίες να ξέρουμε ότι δεν αρκεί μόνο να θεσπίζουμε νομοθεσία, να το μάθουν βεβαίω και τα κράτη-μέλη, κανένα πρόβλημα, να το γνωρίζουν και εκ των προτέρων για, για τις ε, μέλουσες νομοθετικές πράξεις για να ξέρουν και τι του περιμένει. Συμφωνώ, Πέτερ. Αν κρατήσουμε ανοιχτές τις αναφορές θα βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας 100% ναι, σε όλα όσα είπες. Θα μείνει ανοιχτή η αναφορά. Και τώρα. Έχουμε τη βελγική αναφορά. Είναι κάποιος από την Αμβέρσα ο οποίος έχει υποβάλει αυτή την αναφορά όσον αφορά την επιδείνωση της ατμόσφαιρας ε, στο Άμστερνταμ, λέει ο πρόεδρος. Δεν είναι εδώ ο αναφέρον. Ο πρόεδρος εννοεί την Αμβέρσα προφανώς. Έχει το λόγο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Alors, euh, encore une fois, il s'agit d'une pétition assez ancienne qui a fait déjà l'objet. Και σε αυτή την περίπτωση Έχουμε σωρό ανακοινώσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Έχουμε ένα πρόγραμμα όσον αφορά την επέκταση του δικού δικτύου στην Αβέρσα. Αυτό βέβαια έχει συνέπειες ε, στην υγεία, στην ατμόσφαιρα της περιοχής. Όπως ε, προείπα, έχουμε την οδηγία του 2008 ε, που αφορά τα στοιχεία που επιδεινώνουν την ατμόσφαιρα και υπάρχουν οριακές τιμές για διάφορα στοιχεία ε, το PM10 και το διοξίδιο του αζότου. Τα κρατη υποχρεούνται να λάβουν μέτρα για την ατμόσφαιρα. Θα πρέπει τα μέτρα αυτά ε, ούτω ώστε να συγκρατηθεί όσο γίνεται περισσότερο το ξεπέρασμα των οριακών τιμών. Μπορούμε να παρέμβουμε όσον αφορά την υποδομή. Να δούμε δηλαδή ποιε υποδομέ πρόκειται να κάνουν δυσκολότερη τη συμμόρφωση με την νομοθεσία. Ε, Πάντω, ε, περιορισμένο αυτό μπορούμε να κάνουμε, γιατί είναι θέμα αρμοδιότητα των κρατών μελών τελικά. θα πρέπει να βελτιωθεί η, ατμόσφαιρα και να περιοριστούν οι συνέπειε στην ανθρώπινη υγεία. Εμεί παρακολουθούμε το κατά πόσον έχουν μεταφερθεί οι διατάξει τη οδηγία στα διάφορα κράτη-μέλη. Με διάφορε δράσει, με διάφορε πρωτοβουλίε και με την ε, διαδικασία τη ε, παραβίαση του δικαίου. Ήδη αυτό γίνει σε δύο φορές και γίνει για το ε, Βέλγιο, για το PM10 και για το οξύδιο του αζότου και κλείνουμε στάση αναμονής. Περιμένουμε τη συμμόρφωση. Όσον αφορά τώρα την περιοχή της ε, Αμβέρσας, θα πρέπει εδώ να σταθούμε σε μια ιδιοτυπία. Η πόλη αυτή, όσον αφορά το διοξείδιο του αζότου, έχει λάβει κάποια παράταση για να συμμορφωθεί μέχρι το 2015. Σύμφωνα με την οδηγία. Πάντως, ε, τελευταίες εκθέσεις δείχνουν ότι συνεχίζει να υπάρχει υπέρβαση και η περιφέρεια της Φλάνδρας έχει εγκρίνει ένα σχέδιο για την πόλη όσον αφορά την ατμόσφαιρα. Δεκέμβριο του 2017. Ε, λέει ότι βασικά η πηγή του προβλήματος είναι η κυκλοφορία των οχημάτων. Και ε, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα υπάρχει αυτά τα μέτρα, διάφορα μέτρα, όσον αφορά τις οδικές μεταφορές. Προβλέπεται μια ζώνη χαμηλών εκπομπών, η οποία θεσπίστηκε το Φεβρουάριο του 2017. και εκεί θα υπάρχει προοδευτική αύξηση της κυκλοφορίας. Πάντως θεωρείται ότι ε, η παράβαση συνεχίζει να ισχύει. Γιατί οι οριακέ τιμέ που είχαν θεσπιστεί δεν τηρούνται. Οπότε και εμεί θα συνεχίζουμε να παρακολουθούμε με προσοχή την εξέλιξη τη κατάσταση στα πλαίσια τη διαδικασία επί παραβάση, η οποία συνεχίζεται. Professzor Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ και από ό,τι μου αναφέρουν και στην περίπτωση αυτή θα κάνουμε το ίδιο δηλαδή και για την ε, περιοχή αυτή του Βελγίου θα πρέπει να κρατήσουμε αυτή την αναφορά και ούτως ώστε να βελτιώσουμε τις προσπαθίες να διορθωθεί η κατάσταση. Και τώρα, έχουμε τρεις Ιταλικές αναφορές Άννα Τζορμέτα, Ραφαέλε Μπέλετσα και Αντριάννα Πελένη. Έχουν υποβληθεί τρεις αναφορές. Αυτές αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Από ό,τι μου λένε είναι εδώ η κυρία Τζερομέτα, είστε, ναι. Και έχετε το λόγο. Πέντε λεπτά. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τις θέσεις ε, αυτής της ε, ε υπόθεσης που ε, ονομάζεται Τσιταντίνη Περλάρια και ε, βεβαίως θεωρούμε όμως ότι το θέμα αυτό αφορά όλους τους υπογράψαντες εδώ και πολλά χρόνια πολλούς πολίτες και υπάρχουν ε, πάρα πολλά επιχειρήματα που έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα δέχτηκε. Μια που έχουμε αυτή την παράβαση η οποία αφορά την ε, περιοχή της Πάδοβας και γενικότερα την Λομβαρδία. Και τώρα, να σας επισημάνω το πρόβλημα του διοξιδίου του αζότου. Πρόκειται για κάποια ε, κατάσταση που εξελίσσεται, μια παράβαση που εξελίσσεται και η κατάσταση επομένω επήγει. Το 2015 έγινε μια μελέτη από την ε, περιοχή της ε, Ρώμης από Ίδρυμα Επιδημιολογίας. Έγινε μια αξιολόγηση των επιπτώσεων του αζότου του διοξιδίου στη Λομβαρδία και στην Ιταλία. και είπαμε ότι μόνο εκεί κάθε χρόνο στο Μιλάνο έχουμε υπέρβαση του ορίου των 20 μικρογραμμαρίων σύμφωνα με τον ΠΟΕ. Και από την υπέρβαση έχουμε 1650 νεκρούς στην περιοχή του Μιλάνου. Πρόκειται για τα αυτοκίνητα που καίνε ντίζελ. Δεν υπάρχει προστασία ακόμα τώρα και τώρα του κόσμου. Άρα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσφύγει στην διαδικασία που προβλέπεται. Κατ' τα μια που βλέπουμε κυρίως ταξί πάρα πολλά που προκαλούν εκπομπές ιδίω για τα οξύδια του αζότου πολύ παραπάνω τις Βλέπουμε αυτή τη φωτογραφία, τη δορυφορική. 4 Οκτωβρίου, ημερομηνία της δεύτερης ε, Οκτωβρίας για τα οχήματα diesel Euro 3. Ε, προφανώς δεν ισχύουν, δεν, δεν αρκούν τα μέτρα αυτής της κατηγορίας και άρα θα πρέπει τα σχετικά οχήματα να απαγορευτούν, να μην κυκλοφορούν όπως έλεγε προηγουμένως η Επιτροπή, ως ε, πολίτες Ευρωπαίοι ε, ζούμε στη διεθνή μας ζωή το πρόβλημα. Και δημοσιεύθηκε παντού ότι λόγω όλων αυτών των μετρήσεων, όλων αυτών των ε, καταγγελιών πάνω από 300 συμπολιτών μας και επιδημιολόγων ανεγνωρισμένων έχουμε αυτή την παράβαση των 40 μικρογραμμαρίων αζότου ενώ είναι 20 ε, το όριο του ΠΟΕ έχουμε 600 νεκρούς μόνο στην περιφέρεια του Μιλάνου. Ο δε δήμαρχος είπε το 19 τα diesel 1 έως 4, έω θα απαγορευτούν. Αλλά δύο μέρες μετά ο κυβερνήτης, ο Περιφερειάρχης είπε ότι αυτό είναι υπερβολικό. Καταλαβαίνετε επομένω ε, τη σημασία του θέματος. Όπως το εξηγούσε κάποιος λίγο πριν. Θα πρέπει εδώ οι Βρυξέλλες να στείλουν ξεκάθαρο μήνυμα αλληλεγγύης προς τις ε, πόλεις που θέλουν να ληφθούν επιπλέον μέτρα. είναι επομένως πάρα πολύ σημαντικό η διαδικασία για τα οξύδια του αζότου να κινηθεί κατά του Ιταλικού κράτους. Τα οχήματα diesel που είναι πάνω από το όριο να μην κυκλοφορούν στο δρόμο. Να φτιάξουμε ένα ταμείο. Και η πώληση αυτών των οχημάτων. να επιδοτείται. Αυτό θα ωφελήσει τις πόλεις εκείνες. Έτσι θα έχουμε καθαρή ατμόσφαιρα. Και ο κύριος Παρουσίας την μελέτη είπε ότι υπάρχει βελτίωση στο Μιλάνο. Θέλω να σας πω ότι Υπάρχει ένα πρόγραμμα για τη Λομβαρδία, αλλά δεν αρκεί. Είναι πολύ περιορισμένο και σήμερα έχουμε ένα δίκτυο όπου όλες αυτές οι ρηπαντικές ουσίες, κάδμιο, λίθιο κλπ. μετρούνται. Μετρούνται και έχουμε μια περιοχή όπου γίνονται αυτές οι μετρήσεις και υπάρχουν περιορισμοί κυκλοφορίας, αλλά πρόκειται για μια πάρα πολύ, μικρή ζώνη. Μιλάμε για το ένα δέκατο της ζώνης του προβλήματος. Πρόκειται για παραβίαση της σχετικής οδηγίας. Εμείς έχουμε αυτές τις αναφορές για την ατμόσφαιρα, για την απουσία προγραμματισμού. Γι' αυτό σας λέω, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όπως προαναφέρθηκε, ε, είναι ακριβώς όπως είπανε πριν για τα πλοία. Όπως ξέρουμε υπάρχει μια τάση ούτως ώστε να θεσπίζεται στην Μεσόγειο ζώνη χαμηλών εκπομπών. Ε, να έχουμε δύο κατηγορίες ε, ε, ε πλοίων. Να υπάρχουν καύσιμα ε, καθαρά. Άρα θα πρέπει όσο γίνεται ταχύτερα να γενικευθεί η θέσπιση αυτών των ε, ζωνών χαμηλής εκπομπής στην Μεσόγειο. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Και από ό,τι μας λέτε, έχουμε και την κυρία Παλένη εδώ. Και εσείς έχετε πέντε λεπτά. Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε εδώ που εκπροσωπούνται οι πολίτες. Ε, αυτό είναι σύμβολο. Σύμβολο ε, της προστασίας των δικαιωμάτων μας για τα προβλήματα του περιβάλλοντος. Αυτό το υποστέ του περιβάλλοντος ως υγεία μου την είμαι ο πατέρας μου. Και η ανησυχία μας για την ατμόσφαιρα είναι ότι χρειάζεται ε, οξυγόνο και αυτό όμως το, σε όλη την ε, ε, περιοχή της Πάδουα, στην όλη περιοχή της Λομβαρδίας δεν, δεν ισχύει. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω και εγώ και άλλοι συμπολίτες μου ότι θα πρέπει να ισχύσουν οι κανόνες να ληφθεί υπόψη η γεωμορφολογία του τόπου που ζούμε θα πρέπει να ανερθούν τα σχετικά πρότυπα για τις ουσίες που ε, βλάπτουν. Θα πρέπει να δούμε πώς είναι η ρήπανση του ατμόσφαιρας, θα πρέπει να γίνονται καλύτεροι οι, έλεγχοι. Ε, νομίζουμε ότι ο έλεγχος της μόλυνσης αφορά το μέλλον και αυτό επίσης αφορά και τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που μας χτυπάνε. Α, κοιτάξτε εδώ, σας έφερα εδώ αυτά. Ε, Φυτά από το δικό μας δίκτυο που τα καθαρίσαμε γιατί είχαν μεγάλη ρήπανση. Πρόκειται για έναν ε, φορέα εθελοντών και έχουμε εδώ αυτά τα αρώματα που προέρχονται από τους απλούς πολίτες για σας. Barinetti urat kérném az Európai Bizottság képviseletébe. Tessék, parancsoljon. Κύριος Γκασπαρέτη τώρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα σας μιλήσω στα Ιταλικά γιατί σήμερα οι αναφορές μας προέρχονται από Ιταλούς, από αυτούς τους Ιταλικούς φορείς. Είναι πάρα πολύ α, σπουδαίο αυτό το οποίο κάνουν για το χώρο τους. Αν είχαμε τέτοιες επιτροπές εθελοντών που αυθόρμητα οργανώνονται, όπως και στην ε, Λομβαρδία, ε, έτσι θα, θα ταράξουν τα νερά και θα κινητοποιήσουν ακόμα και τα διοικητικά δικαστήρια. Ε, μέσα σε όλη αυτή την αδράνεια που πλήσει την Ιταλία γιατί ε, όλα αυτά είναι λάθη των παλαιότερων κυβερνήσεων. Δυστυχώς η Ιταλία είναι αρνητικός πρωταθλητής όσον αφορά τους πρόορους θανάτους λόγω της βρωμικής ατμόσφαιρας. Είπαμε ότι έχουμε 1.600 θανάτους και παραπάνω κάθε χρόνο. Όλα αυτά τα οποία ανέφερε η κυρία Τζερομέτα ε, είναι πιο συγκρατημένα τα στοιχεία αλλά δυστυχώς έχουμε μετρήσει 60.000 νεκρούς ε, συνολικά. Γι' αυτό λέω ότι το Μηνύο τίμημα είναι πολύ μεγαλύτερο. Όλοι γνωρίζουμε επομένω τι γίνεται, όλα αυτά έχουν μελετηθεί και πολύ σωστά έλεγε η κυρία Τζιρομέτα. Δεν αρκούν αυτά τα οποία γίνονται γιατί όλοι γνωρίζουμε από πλευράς εκπομπών ότι έχουμε όλα αυτά τα σωματίδια που εκπέμπονται από τα αυτοκίνητα και των προδιαγραφών Euro 5. και στην Ιταλία υπάρχουν περιορισμοί στην κυκλοφορία ε, για τα Euro 2 και Euro 3. Δεν γίνονται αρκετά. Ξέρετε τις εργάσιμες μέρες υπάρχουν άδειες σε 12.000 οδηγούς που εξαιρούνται από τα μέτρα να δείξουμε τι γίνεται και στην Γερμανία. Ακόμα και πέρα από 80 πόλεις που έχουν πιο σοβαρά ε, μέτρα. Μια που είστε πολιτικό όργανο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ότι οι πολλοί από, τη, ε, από όργανο προσπαθήσει να καθυστερήσουν, να φρενώνουν αυτά τα μέτρα. Ε, είπαμε ότι θα πρέπει να μελετηθούν τα μέτρα τα οποία όμως δεν έχουν αποφέρει αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε αλλακτική λύση. Και γι' αυτό προσέφηκε στην δικαιοσύνη κατά της Ιταλίας. Τώρα για την ε, Λομβαρδία. Ε, Λαμβάνει την υπόψη και το τι έχει γίνει με Βουλγαρία και Ρουμανία. Οι δικαιολογίε που προτάθηκαν ήταν οικονομικές ε, δυσκολίες. Φτώχεμα δεν ισχύει αυτό για την ε, Ιταλία. Μιλούμε από πλευράς ΑΕΠ για τις πιο πλούσιες. Το ΑΕΠ είναι τόσο υψηλό που τελικά το θέμα είναι πολιτικής επιλογής. Πρόκειται περί μεγάλης οικονομίας που θα γινόταν εάν προστατεύονταν η υγεία των πολιτών. Αυτό είναι καθήκον για την πολιτική τάξη. Είναι επένδυση σε οικονομικούς όρους. για κάθε μία ώρα προστασίας έχουμε 12 ώρες παραγωγικές. Αυτό αφορά τη διοίκηση της επιχειρήσης όλους. Γιατί ακριβώς έχουμε απουσιασμό από αυτούς που αρρωσταίνουν. Επομένω, πρέπει κάτι να γίνει και από οικονομικής πλευράς. Και κλείνω τονίζοντας ότι είχαμε και τα προηγούμενα Πολωνίας Βουλγαρίας και λέμε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα έχει τα ίδια κριτήρια. Ότι δηλαδή τα ληφθέντα μέτρα δεν είναι αρκετά. Ότι έχουμε επιδείνωση της κατάστασης σχέση με το παρελθόν. η Βενετία. Δεν έχει αυτοκίνητα. Δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα, είναι όλα πεζόδρομοι. Εκεί. Έχουμε όπως στο Μιλάνο και στο Τωρίνο εθαλομίχλη. Σε όλη τη Λομβαρδία ισχύει αυτό. Γιατί, πάντα λέμε ότι είναι θέμα των οδικών μεταφορών. Και βέβαια βλέπουμε ότι αν δοθεί προτεραιότητα στην κυκλοφορία των πεζών και όχι των αυτοκινήτων, αυτό μπορεί να βοηθήσει. Πάντω θα μπορούσαν να δοθούν λύσεις εκ πέραν του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και στα εθνικά δικαστήρια. Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην κυρία Εύη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους αναφέροντες και την Επιτροπή. Μας περιγράψει την κατάσταση που όλο ένα και περισσότερο πιέζει θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. είναι αφόρητο να συνεχίζουμε να ακούμε για το, όλα αυτά τα στοιχεία. Πόσοι πρόωρα πεθαίνουν. Πόσα χρόνια χάνονται από τη ζωή ενός ανθρώπου. Πένθος. Θλιβερό και αυτό το τι γίνεται με τους θανάτους των ανηλίκων στην Ιταλία που είναι πολύ χειρότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Μιλάμε για 90.000 τέτοιους πρόορους θανάτους. 440.000 είναι το σύνολο της Ευρώπης. άρα θα πρέπει κάτι να κάνει η Ιταλία να λύσει το πρόβλημα που τραβάει τόσα χρόνια. Δεκαετίες. Κανείς δεν έκανε μέχρι σήμερα. Τίποτα δεν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Να, και θέλουν να τα κουκουλώσουν τώρα. να συζητούμε ακριβώς τη συγκεκριμένη περιοχή, Λομβαρδία, Πεδεμόντιο, Εμίλια, Ρωμάνια, ε, πρόκειται για κάποιες περιοχές που δεν έχουν αξιόπιστα μέτρα για να προστατεύσουν την ατμόσφαιρα. Συμφωνώ με την κυρία Τζιρομέτα ότι φταίνε τα diesel Euro 3 αλλά η απαγόρευσή τους δεν αρκεί γιατί είναι πάρα πολλά τα ντίζελ που ρηπαίνουν και κυκλοφορούν στις πόλεις μας. Υπερβαίνουν τις τιμές, τα όρια. Μα έτσι κι αλλιώς τα πιστοποιητικά και αυτά που προβλέπονται βγαίνουν από βγαίνουν σε εργαστήρια στην πράξη. Οι εκπομπές όπως και στο Dieselgate είναι 20 φορές πιο μεγάλες. θα έπρεπε στην ώρα τους να έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά. Αποτελεσματικά είναι τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν. Ή μάλλον θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά και θα πρέπει να υπάρξει απαγόρευση κυκλοφορίας. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να μελετηθούν το νωρίτερο. Ε, πολλές φορές ξεχνάμε το retrofitting. Το τι μπορούμε να κάνουμε για τα αυτοκίνητα που ήδη κυκλοφορούν. Υπάρχουν λύσεις. Στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας. Που μπορεί να ωφελήσει σε περίπτωση που πρέπει να βγει από την κυκλοφορία το αυτοκίνητο. Ναι, οι φιλόδοξοι νόμοι χρειάζονται. Και να επιβληθεί στην βιομηχανία τι θα πρέπει να παράγουν, τι θα πρέπει να ρίχνουν στην αγορά. Έτσι θα πρέπει να είναι ναι, οι κανόνες για τις εκπομπές των οχηματών. Όπως και οι προηγούμενες αναφορές να μείνουν και αυτές ανοιχτές. Έτσι θα δείξουμε τι κατεύθυνση θέλουμε να πάρουν τα πράγματα. Θα πρέπει να πέσει το βάρος της ε, δημόσιας μεταφορές. στη δική μου περιοχή, στη Λομβαρδία. Έγιναν επενδύσεις, έγιναν υποδομές. Αυτοκινητόδρομοι, δρόμοι, εμπορικά, ε, εμπορικά κέντρα. Και όλα αυτά όμως οδηγούν σε περισσότερη ρήπανση. Να μείνουν ανοιχτές οι αναφορές και έτσι να πάρει η πολιτική μας αυτή την ε, κατεύθυνση. Και κατόπιν της ε, προσφυγής στη δικαιοσύνη θα πρέπει οι περιοχές που έχουν παραβεί το νόμο να υποστούν πρόστιμο. Βάλει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ συμφωνώ με τους αναφέροντες και με την Ελεονόρα Εύη. Και εγώ προέρχομαι από εκεί, από τη Λομβαρδία, κοντά στο Μιλάνο. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα όσον αφορά την ε, ατμόσφαιρα. Από τεφρώσεις, αυτοκίνητα, πάρα πολλές είναι οι αιτίες. Ακόμα και η θέρμανση σπιτιών και δημοσίων κτηρίων. Δεν είναι τα πράγματα όπως θα έπρεπε για να τηρηθούν τα πρότυπα, οι οριακές τιμές τέλος πάντων. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθήσει γιατί έχουμε ε, το, το, δημόσιο κορβανά που θα έπρεπε να εφίσταται καλύτερη διαχείριση εκεί πέρα. Είπαμε, όταν ε, ενεργοποιείται η θέρμανση, κορυφώνεται η ρήπανση. Οι καυστήρες είναι το πρόβλημα, οι λέβητες. Α αξιοποιηθούν καλύτερα οι πόροι τη περιφερειακή ανάπτυξης. Αν κάτι άλλο, στον την Τράπεζα Επενδύσεων, που ξέρουμε ότι είναι ανεξάρτητη αρχή, αλλά κατά τη γνώμη μου, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να πιέσει περισσότερο την ΕΤΕ. Γιατί πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια έχουμε εγγυήσεις χρηματοδοτήσεων ή χρηματοδοτήσεις στον ιδιωτικό τομέα που χρηματοδότησαν τελικά κάποια απειρχαιωμένα έργα. Έχουν ευνοήσει το αυτοκίνητο. Δεν έχουν πάει αυτά τα χρήματα σε πιο καθαρές υποδομές. Άρα, η ΕΤΕ θα πρέπει να κάνει τη δουλειά για την αποστολή της μπορεί να δώσει μια προσθεμένη αξία όσον αφορά τη βελτίωση ε, της πολιτικής του περιβάλλοντος. τα έχει πει αυτά η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού και Προϋπολογισμού. Με μεγαλύτερη επιμέλεια θα πρέπει η ΕΤΕ να χρηματοδοτεί με εκατομμύρια αυτά τα έργα στην Λομβαρδία. Γενικότερα στη Βόρεια Ιταλία. Οπωσδήποτε να μείνουν ανοιχτές αυτέ οι αναφορές. Να συνεχίσουμε να πιέζουμε. Με ό,τι μπορούμε να πιέσουμε όποιες αρχές πρέπει και ευρωπαϊκές. Και έτσι οι επενδύσεις που γίνονται να είναι καλύτερες. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Επίσης, να ευχαριστούμε και τον Μάριο Γκασπαρινέτη. Τα μας τα είπε πολύ ολοκληρωμένα. Συμφωνούμε μαζί σας. Είμαστε στο πλευρό σας. Ευχαριστούμε για τις ε, απόψεις που μας αναλύσατε. Ευχαριστούμε τους αναφέροντες και ευχαριστούμε που αναδείξατε αυτό το θέμα. Αμήνων ανοιχτές οι αναφορές και θα συνεχίσουμε τον διάλογο θα συνεχίσει να τρέχει η διαδικασία επί παραβάση κατά της Ιταλίας κυρία θέλετε το λόγο πάλι μήπως μπορούμε να απευθύνουμε στην περιφέρεια αυτήν αυτές μάλλον Εμίλια Ρωμάνια Πεδεμόντιο Λομβαρδία που αναφέρονται εδώ να τους απευθύνουμε να τους στείλουμε τέλος πάντων αυτή τη μελέτη που αναλύσαμε σήμερα. Α, και στην περιφέρεια της Βενετίας επίσης. Ο Πρόεδρος. Πολύ σωστή η πρότασή σας. Συμφωνούν οι αναφέροντες. Με αυτά τα οποία συστήνουμε. Ναι. να μείνουν ανοιχτέ οι αναφορέ. Και θα στείλουμε στις περιφέρειες που εμπλέκονται την μελέτη που σήμερα παρουσιάσαμε εδώ. Και βέβαια βοηθούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο δικό της έργο. Γκασπάρη, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε πάλι το λόγο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κάνετε αυτό, διότι η Κομισιόν, όπως γνωρίζετε, όταν επεξεργάζεται διαδικασίες επί παραβάση, μπορεί να μιλήσει μόνο, μόνο με τα κράτη-μέλη. Αυτό για το οποίο μιλάμε τώρα είναι καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που μόνο εν μέρη εναπόκειται στις εθνικές κυβερνήσεις. Γιατί στην Ιταλία τα ζητήματα που σχετίζονται με την ποιότητα του αέρα είναι αρμοδιότητα των περιφερειών. Σε κάποιες περιφέρειες λοιπόν υπάρχουν βελτιώσεις, έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Διότι ε, η κάθε ε, τοπική αυτοδιοίκηση, κάθε αρχή, τοπική αρχή μπορεί να έχει την πολιτική βούληση για να λάβει μέτρα ή όχι. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, και πολύ χρήσιμο αν ακολουθήσετε αυτή την οδό. Αν δηλαδή ε, μπορέσει να διαδοθεί και μέσω των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης το τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ποιότητα του αέρα στην Ιταλία. Να προσθέσω ότι στην αναφορά μας αρχικώς ασχοληθήκαμε και με το ζήτημα του σχεδιασμού για την ποιότητα του αέρα. Προφανώς το, το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό στην κοιλάδα του Πάδου, αλλά όχι μόνο. Μιλάμε για το Λάτσιο, την Καμπανία, πολλές άλλες περιοχές λοιπόν πλήττονται και αυτές από την πολύ χαμηλή ποιότητα του αέρα και γι' αυτό θα ήταν πολύ θετικό να λάβουν και εκείνες την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ναι, ναι, πρόκειται να απευθύνουμε επιστολές στις ε, αντίστοιχες ε, περιφέρειες της και επίσης θα στείλουμε και τη μελέτη που εξετάσαμε το πρωί. Θα μείνουν ανοιχτέ οι αναφορέ και επίση στηρίζουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι προσπαθίε τη. Εντάξει, ναι, ωραία. Για σήμερα έχουμε την ε, τελευταία αναφορά. Πρόκειται το Σαμόλ Μαρτίν Σόσα. Έχει υποβάλει μια αναφορά από την Ισπανία. Χουάν Γκαρσία Βισέντε. Είστε εδώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πάνω από 14.000 νεκρούς στην Ευρώπη και στην Ισπανία. Και έχουμε μόνο ένα τμήμα που αφορά το όζον. Και ιδίως αυτό αφορά το κέντρο, το νότο της Ισπανίας, τις ακτές της Μεσογείου. Οπότε τώρα βλέπουμε ότι διακόπτει ο Πρόεδρος Ξέρετε, έτσι όπως τα λέτε, δεν υπάρχει περίπτωση να σας μεταφράσουν. Μπορείτε να τα λέτε πιο αργά. Έχουμε το άρθρο 3 τη Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο ορίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και το άρθρο 17 αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την, τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικτύου. Έχουμε την οδηγία 2008-50 που έχει σχέση με την ποιότητα της ατμόσφαιρας ε, που πρέπει να είναι πιο καθαρή στην Ευρώπη και στο σημείο 18 λέει ότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, κάποια προγράμματα για την ποιότητα της ατμόσφαιρας, για τις ζώνες, για τις περιοχές όπου ε, δεν ισχύουν οι τιμές στόχοι και αυτά προβλεπούνται στο άρθρο 23 της οδηγίας που είπαμε. Παρ' όλα αυτά έχουμε μία ντουζίνα από ισπανικές περιφέρειες 250.000 τετραγωνικών και 20 εκατομμυρίων κατοίκων που δεν τηρούν αυτές οι ωρακές τιμές. Και επίσης εδώ έχουμε α, τις αρμόδιες αρχές που δεν έχουν κάνει ό,τι πρέπει και ό,τι λέει η Οδηγία 2050. Ε, πρόκειται για τις περιφέρειες Ανταλουσίας, Αραγωνίας, Βαλεαρίδων, Καστήλες, Καστήλες Λεών, Καταλανίας, Βαλεντίνη, Εξτρεμαδούρα, Μούρθια, Μαδρίτη, Ναβάρα και χώρα των Βάσκων. Πρόκειται για πάρα πολύ βαριά αμέλεια πλευρά ε, τη διοίκησης που παραβλάπτει ε, την υγεία, την ε, γεωργία, τα δάση και γι' αυτό το λόγο ε, οι οικολόγοι σε δράση, όπως λέγεται αυτή η, η οργάνωση, απευθύνει Ευρωπαϊκή τον Ιούλιο του 2016 και ζήτησε να γίνει διαδικασία παραβάση όσον αφορά το βασίλειο της Ισπανίας και έτσι θα πρέπει το κράτος να εκπονήσει κάποια τέτοια προγράμματα για προστασία της ατμόσφαιρας όπως ορίζει το δίκαιο. Παρ' όλα αυτά, ε, η καταγγελία μας μπήκε στο αρχείο τον Αύγουστο και είπαν ότι η τήρηση των στόχων για το α, όζον έχει γίνει. Είναι μάλλον περίπλοκη η υπόθεση, είπε, γιατί πρόκειται για δευτερογενή πηγή μόλυνσης. Γι' αυτό και εμείς απευθυνθήκαμε στο Κοινοβούλιο. Θέλουμε να πιέσετε την Επιτροπή, ούτω ώστε να τηρήσει την υποχρέωσή της. Και στην ε, απάντηση του Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε στο Κοινοβούλιο ότι αποφάσισε να επικεντρώσει τις προσπάθειές της όσον αφορά την τήρηση των ε, διατάξεων ε, ποιότητας ατμόσφαιρας και να δοθεί προτεραιότητα σε αυτά τα προβλήματα. Να δούμε τι γίνεται με τα διάφορα μόρια και σωματίδια που αιωρούνται ε, το PM10, το διοξίδιο του αζότου, να, να καταβληθούν προσπάθειες που να δίνουν, να αποδίδουν τη σημασία που πρέπει. Και θα πρέπει να δούμε το ότι πρέπει να πιεστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απευθύνει τη διαδικασία παραβάσης προς την Ισπανία που δεν κάνει ό,τι πρέπει. Οι οικολόγοι σε δράση πιστεύουν ότι χρειάζεται να υπάρξει έλεγχος όσον αφορά την τήρηση αυτών των υποχρεώσεων των υποχρεώσεων για προστασία της ατμόσφαιρας. Πρόκειται για δεκάδες εκατομμυρίων Ευρωπαίων που παραβλάπτονται γιατί συστηματικά παραβιάζονται οι οριακές τιμές που αφορούν ε, την ε, φύση, τα φυτά, την υγεία. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση στη μεγαλύτερο τμήμα της Ισπανίας. Ε, αυτό σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να πιέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει την εφαρμογή του δικαίου. Έτσι, θα πρέπει να συγκρατηθεί η ρήπανση από το όζον. Αυτό να γίνει το συντομότερο. Ακριβώς όπως λέει η πρόσφατη σύσταση του ελεγκτικού συνεδρίου ο πρόεδρος. Να δώσουμε τον λόγο στην εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και τον αναφέροντα για τα θέματα που έθεσε σχετικά με την ποιότητα του αέρα στην Ισπανία καθώς και για το γεγονός ότι αναδεικνύει μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα η Κομισιόν επισημαίνει ότι ο περίπλοκος μηχανισμός σχηματισμού του όζοντος στην ατμόσφαιρα δεν είναι ο μόνος λόγος που αιτιολογεί την, τη διαδικασία επιπαραβάσης που έχει ξεκινήσει η Κομισιόν. Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στις υπερβάσεις ε, διοξιδίων του ε, αζότου και τα ε, μικροσωματίδια όσον αφορά τις διαδικασίες επιπαραβάση. Ωστόσο, ε, περιμένουμε αυτές τις διαδικασίες, ιδίως όσον εκείνες που αφορούν το διοξίδιο του αζότου, να βελτιώσουν και την κατάσταση του όζοντος, καθώς ε, το διοξίδιο του αζότου είναι πρόδρομη ουσία για, το σχηματισμό όζοντος στην ατμόσφαιρα. Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι τα νέα, ε, η νέα οδηγία για τα εθνικά όρια επίσης αναμένεται να βελτιώσει την κατάσταση όσον αφορά την συγκέντρωση του όζοντος, διότι η οδηγία αυτή ε, καθορίζει συγκεκριμένε δεσμεύσει μείωση των, των εκπομπών για, ε, για πρόδρομε ουσίε όπω είναι πτυτικέ ενώσει κτλ. Οξύδια του αζότου κτλ. Ωστόσο, με την επιφύλαξη αυτών των διαδικασιών επί παραβάση, η Κομισιόν επίση ε, βρίσκεται σε επαφή με την Ισπανία και συζητά ζητήματα ε, ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και του όζοντος και για την αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων μέσω άλλων ε, μηχανισμών. Υπάρχει ο διάλογος για τον καθαρό αέρα, για παράδειγμα. Αυτός ε, διεξάγεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Μαδρίτη, ο διάλογος αυτός, και είναι ένα προστηρητικό πρόγραμμα το οποίο έχει σχεδιαστεί προκειμένου να αξιολογείται να αξιολογούνται τα πλέον πιεστικά προβλήματα που αφορούν στην ποιότητα του αέρα στα κράτη-μέλη και δίνει τη δυνατότητα να συζητηθούν τα πλέον αποτελεσματικά μέτρα και πολιτικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Μια άλλη διαδικασία που μπορούμε να προτείνουμε είναι ένα εργαστήριο συγκεκριμένα για το όζον που θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο στη Μαδρίτη και που θα διοργανωθεί από τις Ισπανικές Αρχές σε συνεργασία με τις Γαλλικές Αρχές καθώς και με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο της, του μηχανισμού ε, ομοτήμων για την αναθεώρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής. Επίσης, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση που αφορά τον, την ποιότητα του αέρα στην Ισπανία και αυτό περιλαμβάνει και την πλήρη αξιολόγηση των δεδομένων που, θα λάβ, που λάβαμε για το 2017 από την Ισπανία στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστώ. Κύριε Βαλίνη, έχει το λόγο, λέει ο Πρόεδρος. Πρώτα-πρώτα ευχαριστούμε τους αναφέροντες. Η ρήπανση από το ακριβώς, όπως και από κάθε ρηπαντική πηγή, αποτελεί προτεραιότητα ως αντικείμενο αντιμετώπισης γιατί οι συνέπειες είναι όλοι αυτοί θάνατοι. Μιλούμε για χιλιάδες ανθρώπων που κάθε χρόνο πεθαίνουν από την ρήπανση. Είναι ό,τι χειρότερο για το περιβάλλον. Με ανησυχεί πάρα πολύ η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Ακούσαμε τι γίνεται και στην Ιταλία. για την Ιταλία εντάξει, ήταν κάπως πιο φασιστική, αλλά κοιτάξτε, θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι να γίνει διαδικασία υπερβάση για την Ισπανία, μια που δεν υπάρχουν ε, ε, μέτρα για βελτίωση της ατμόσφαιρας στην Ισπανία, όποτε έχουμε υπέρβαση των τιμών για το όζωνα, σύμφωνα με την οδηγία, είπαν ότι δεν είναι το πιο σωστό ε, μέτρο. Όμως επαναλαμβάνει η Επιτροπή ότι θέλει ατμόσφαιρα πιο καθαρή στην Ευρώπη. Θα συνεχίζει να μελετά τι μηχανισμοί υπάρχουν ούτω ώστε να μην υπάρχει συγκέντρωση του οζόνου του όζοντο, συγγνώμη, οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε χρειάζονται κάποια προγράμματα δράσης όπου χρειάζεται. Όπου χρειάζονται προγράμματα, ούτως ώστε να ισχύσουν οι οριακέ τιμέ. Μα όλα αυτά είναι αντίφαση, είναι η ίδια η αντίφαση. Μα ανησυχούμε γιατί υπάρχει υπέρβαση των τιμών και δεν εφαρμόζεται η οδηγία, αλλά από την άλλη μεριά δεν θα κάνουμε τίποτα, θα κάνουμε αυτό το εργαστήρι. Μα τι να κάνει το εργαστήρι, τι μέτρα να λάβει για την ρήπανση αυτή, η απάντηση αυτή. Τι να σας πω, ειλικρινά δεν την καταλαβαίνω. Πρόκειται για κοροϊδία, κοροϊδία προς όλους αντίφαση. Επίσης λέμε ότι είναι δεδομένη αυτή η μελέτη. Γιατί έχουμε διαδικασία παραβάση κατά 16 κρατών ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ακριβώς για το ζήτημα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης και υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το θέμα αυτό της προσφυγής στο δικαστήριο. Να δοθεί ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα για να συμμορφωθεί η Ισπανία. Προτείνω στην Επιτροπή μας να κρατήσει ανοιχτή την αναφορά και να συνεχιστεί η διερεύνηση της υπόθεσης. Να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ισπανικές αρχές τι απάντησαν, τι επιχειρήματα προέταξαν. Θα πρέπει η Ισπανία να λάβει μέτρα και να μας πει τώρα τι κάνει, γιατί τώρα θα πρέπει να συγκρατηθεί η ρήπανση. Μαρτσελίση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε αυτή την οργάνωση τους ε, οικολόγους που έχουν αναλάβει δράση. Ξέρουμε τι γίνεται σε χώρες όπως η Ισπανία. Ξέρουμε ότι σκοτώνει η ρήπανση. Μα το λένε τα νούμερα. Δεκάδες χιλιάδων είναι οι νεκροί. Και είπαμε 1600 μόνο στην Ισπανία. Μιλάμε για το 44% της έκτασης, το 30% των Ισπανών παίρνουν μέσω της αναπνοής όλο αυτό το όζον. Και η οδηγία 50 του 8 τα λέει. Θα πρέπει να επιθυμιστεί το ότι άλλοι λαμβάνουν μέτρα, άλλοι όχι. Έτσι θα χαρακτηριστεί τη στρατηγική μας. Να κάνουμε κάτι για τις περιφέρειες που δεν κάνουν το καθήκον τους. Μιλάμε για κράτος το οποίο δεν αντιδρά. Μαδρίτη, Βαρκελόνη, ε, θα πρέπει όλες οι πόλεις να κάνουν ό,τι μπορούν για να σταματήσει να πεθαίνει ο κόσμος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα στην Ισπανία. Αναγνωρίζει ότι παραβιάζεται η οδηγία. Αλλά η απάντηση είναι ανεπαρκής. Εμείς τι κάνουμε τώρα. Αφήνουμε ανοιχτή την αναφορά και ζητούμε περισσότερη ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ανεπαρκής η απάντησή σας. Συμπαθάτε μας. Και απευθύνουμε επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ισπανίας. Η κυβέρνηση έφτιαξε αυτό το Υπουργείο που το λέει Υπουργείο οικολογική μετάβασης. Ωραίο το όνομα, αλλά για να μας πούν τι είναι, διακοσμητικό ή θέλουν να έχουν πολιτική που να ανταποκρίνεται, που να αντιστοιχεί στο όνομα του Υπουργείου. Να συγκρατηθεί αυτή η ρήπανση. Μα είναι δυνατόν να μην μπορούμε να, ξεκαθαρίσουν τι θέλουν. Μια πολιτική που σώζει ζωές ή που σκοτώνει. Ο κύριος Γιάρ. Συνάδελφοι, θέλω να προστατεύσω λίγο την Κομισιόν σε αυτό το θέμα, διότι η Κομισιόν το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να αντικατοπτρίζει ποια είναι η κατάσταση και να μας την περιγράφει. Η κατάσταση είναι αυτή που είναι. Φυσικά, ε, πολλές φορές ε, με ρωτάνε θέλετε περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη. Εγώ απαντώ, θέλω Ευρώπη στην οποία οι νόμοι που θεσπίζουμε θα εφαρμόζονται. Στη Γερμανία μάλιστα ε, υπάρχουν κάποιες χώρε. Ε, υπάρχουν πόλεις μάλλον που επέρονται ότι έχουν πολύ καλό αέρα, πολύ καλή ποιότητα του αέρα. Και άμα κοιτάξει λίγο καλύτερα κανείς τις περιπτώσεις αυτών των πόλεων, απλώς είναι τυχερές λόγω της γεωγραφικής τους θέσης. Ε, φαίνεται ότι για άλλη μια φορά δεν έγινε καλή δουλειά όταν θεσπίστηκε η σχετική νομοθεσία. Γιατί είπαμε εντάξει, okay, ας βάλουμε αυτές τις οριακές τιμές και θα τις, ε, θα τις επιτύχουμε και χωρίς να έχει εκτιμηθεί σε βάθος αν πράγματι υπήρχε δυνατότητα να, γίνει, ε, να τηρηθούν όλα αυτά τα όρια. Νομίζω ότι όλα αυτά που έχουμε συζητήσει σήμερα στην πρωινή μα συνεδρίαση πρέπει να τεθούν υπόψη τη Επιτροπή Περιβάλλοντο. Γιατί μπορούμε να καθόμαστε να παραπονιόμαστε, αλλά αυτό που μα ενδιαφέρει στην πραγματικότητα είναι να σημειωθεί πρόοδο. Και πρόοδο δεν μπορεί να γίνει μέσα τρία λεπτά που θα εξετάσουμε κάθε ε, αναφορά. Όμως μπορούμε να δώσουμε την αίσθηση στους αναφέροντες ότι πραγματικά υπάρχει βούληση από τη δική μας πλευρά να βελτιωθεί η κατάσταση και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία μας με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, φυσικά ε, η επαφή μας με τις ε, υπηρεσίες, τη της Κομισιόν και αλήθεια σα λέω ε, υπάρχουν, υπάρχουν πάρα, πάρα, διαστάσεις του θέματος ε, να ε, ε, εκνευρίζομαι και με τι αποφάσει που παίρνονται στη Γερμανία. Ε, απαγορεύουμε τα οχήματα diesel, ναι, αλλά με τα χιλιάδες άνθρωποι που, ασχολούνται στα συνεργεία, που απασχολούνται στα συνεργεία, για παράδειγμα, τι θα κάνουν. το πρόβλημα, λοιπόν, είναι πρώτον, να αναπτυχθούν μέτρα, να ληφθούν μέτρα πολύπλευρα, πολύμορφα, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τι ιδιαίτερότητε του κάθε κράτου μέλους, τη κάθε πόλης, τη κάθε περιφέρεια, Αυτά όμω θα πρέπει να συνεκτιμώνται στη φάση τη θέσπιση και του καθορισμού των ανώτητων ορίων προκειμένου όλα αυτά να μπορούν στη συνέχεια και να εφαρμόζονται. Ζήτημα δεν είναι και ζητούμενο δεν είναι μόνο να θεσπίζουμε νομοθεσία αλλά να είμαστε και βέβαιοι ότι όλη αυτή η νομοθεσία θα μπορεί και να εφαρμοστεί στην πράξη. Ευχαριστώ πολύ κύριε και κύριοι. Ε, θα μείνει ανοιχτή η αναφορά και πρόκειται να απευθύνουμε αυτή την ε, ε, επιστολή όπως προτείνει ο κ. Μαρθελέζη προς το αρμοδίο Υπουργείο. Και κατά αυτόν τον τρόπο κύριε ε, Γιάρ θα βοηθήσουμε και την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αλλά τώρα να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Βιθέντε για δύο λεπτά. Είστε ο αναφέρον, θέλετε ξανά το λόγο. Ευχαριστώ που μας καλέσατε. Ναι, ναι, θα πρέπει να έχει αυτή αφορά γιατί αυτό θα βοηθήσει να βελτιωθεί η ατμόσφαιρα. Είπαμε ότι θίγονται πάρα πολλοί Ισπανικοί. Ε, συγγνώμη, πάρα πολλοί Ισπανοί και μεγάλο τμήμα της χώρας κυρίως κοντά στη Μεσόγειο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει ξανά το λόγο. Ευχαριστούμε. Θέλουμε να δώσουμε κάποιε περαιτέρω εξηγήσει όσον αφορά τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε σε σχέση με τι διαδικασίε επί παραβάση. Πολύ σύντομα, πρέπει να σημειωθεί ότι το όζον αφενό και τα σωματίδια και το διεξίδιο του αζότου αφετέρου δεν υπόκεινται στην ίδια ακριβώ ε, μεταχείριση ε, στην οδηγία για την ε, ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και μάλιστα υπάρχουν διαφορετικές υποχρεώσεις των κρατών μελών. Συγκεκριμένα για το όζον περιγράφει η οδηγία μια τιμή στόχο που μπορεί να επιτευχθεί μέσω μέτρων που δεν επιφέρουν δυσανάλογο κόστος που δεν είναι το ίδιο με τον υπήρχε μια οριακή τιμή, η οποία θα έπρεπε να τηρηθεί υποχρεωτικός. Επιπλέον, αν κάποια ε, τιμή στόχος παραβιαστεί, όπως για παράδειγμα στο παράδειγμα, του, του όζοντος, τότε διαδικασίες επιπαραβάση, τότε μάλλον μέτρα λαμβάνονται μόνο εφόσον κρυ, κρυθούν κατάλληλα από τα κράτη-μέλη. Άρα η Κομισιόν θεωρεί ότι οι διαδικασίες επιπαραβάση για την αντιμετώπιση ουσιών πρόδρομων του όζοντος, ε, όπου υπάρχουν πολύ αυστηρές διατάξεις, θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο γόνιμες σε τελική ανάλυση και που θα ωφελούσαν και το, την ε, συγκέντρωση όζοντος στην ατμόσφαιρα. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι αρνούμαστε ότι υπάρχει πρόβλημα με το όζον. Φυσικά και υπάρχει και είναι πολύ σοβαρό. Και είναι και πολύ περίπλοκο. Και γι' αυτό το λόγο το εργαλείο peer-to-peer -peer ε, to peer ειναι που θα χρησιμοποιηθεί στο εργαστήριο είναι πάρα πολύ σημαντικό ώστε να μπορούν οι προγνώμονε των κρατών μελών να ανταλλάξουν απόψει και γνώσει σχετικά με την εμπειρία που έχουν συλλέξει κατά την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματο. Δεν μπορεί να πει κανεί ότι το ένα μέτρο ή το άλλο θα οδηγήσει σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα και ότι αυτό θα γίνει μάλιστα και αναγκαστικά και σίγουρα, γιατί καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα, ε, μια ουσία που δημιουργείται στο, ε, στην ατμόσφαιρα από την αντίδραση τη χημική κάποιων ουσιών με την ηλιακή ακτινοβολία. Παρ' όλα αυτά δουλεύουμε σε πολλά μέτωπα, η Κομισιόν κάνει, παίρνει πολλά μέτρα θα συνεχίσουμε τις επαφές μας με τις ισπανικέ αρχέ, θα αναλύσουμε και τα δεδομένα που μας στείλαν για το 2017 και από εκεί και πέρα θα καθορίσουμε και τα επόμενα βήματά μας. Ε, σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Οπότε αποφασίζουμε να μην ανοιχτεί η αναφορά και περιμένουμε την απάντηση επίσης ε, του αρμοδίου Ισπανικού Υπουργείου ε, αυτά για σήμερα το πρωί. Σας ευχαριστώ. Και συνεχίσουμε στις 2.30. Στις με τους φίλους από την ε, Γερμανία. Καλή όρεξη σε όλους.